Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen im Europäischen Parlament. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τη διακοινοβουλευτική ε, διάσκεψη καλωσορίζω όλους ιδιαίτερους τους συναδέλφους ε, των κρατών μελών. 20 εκπροσώπους έχουμε σήμερα παρόντες από τα διάφορα κρατημέλη. Ελπίζω να λειτουργεί σωστά και καλά η μετάφραση, να μας ακούτε σε όλες τις γλώσσες, να μπορέσουμε να μιλήσουμε τη γλώσσα μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως ε, σύνθημα ενωμένη στην ε, πολυμορφία. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί τη βάση μιας καλής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή η διακοινοβουλευτική συνεργασία, η ανταλλαγή απόψεων ε, με τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό χαίρομαι που ήρθατε σήμερα να συζητήσουμε θέματα ελέγχου του προπολογισμού χρηστής διαχείρισης ε, δημοσίων κονδυλίων. Έχουμε μία μερίσια διάταξη που στο πρώτο τμήμα της εξετάζει την έκθεση της κυρίας Βαϊκιένε, ελπίζω να μην έκανα λάθος το όνομά σας, που είναι η πρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου προπολογισμό στη ΣΕΙΜΑ, στη Βουλή της ε, Λιθωνικής Δημοκρατίας. Και ε, από την άλλη έχουμε τον κύριο Ντασίλβα Καλδέρα που είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Είναι δημόσια η συνεδρίαση με τις αντίστοιχες γλώσσες ε, και ε, μεταδίδεται και στο διαδίκτυο. Αν συμφωνείτε με την ημέντησια διάταξη που σας έχει υποβληθεί, ε, την εγκρίνουμε. Και βέβαια σε κάθε σημείο έχουμε και συζήτηση. Δεν βλέπω να επιθυμεί κανείς τροποποίηση της ημέρησης διάταξης και προτείνω να προχωρήσουμε έτσι. Εισαγωγικά θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στη σημασία του ελέγχου του προϋπολογισμού. Είμαστε ακράδοντα πεπισμένοι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ακριβώς ε, όταν το ταμείο είναι μείον και υπάρχουν δημοσιονομικά προβλήματα ε, στον προπολογισμό των κρατών αλλά και των περιφερειών και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι όλο και πιο δύσκολο το έργο μας και το καθήκον να φροντίζουμε ε, τα χρήματα των φορολογουμένων να πιάνουν τόπο. Όχι απλώς δηλαδή να δαπανώνται νομότυπα, αλλά και αποτελεσματικά και να επιτυχάνονται οι επιθυμητοί στόχοι με όσο γίνεται λιγότερους πόρους. Ε, να δαπανώνται σωστά, ε, νόμιμα και να πιάνουν τόπο, επαναλαμβάνω. Και εδώ στο Κοινοβούλιο στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού έχουμε μια ε, πολύ ε, ενδιαφέρουσα συζήτηση που αρχίσαμε πριν από λίγο καιρό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο γιατί θεωρούμε ότι στο μέλλον ο προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει ε, να είναι στραμμένος και προσανατολισμένος προς τις επιδόσεις performance-based λέγεται αυτό στα αγγλικά, ε, είναι μια αλλαγή στο σχεδιασμό και θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να ρίζουν στόχους, πολιτικούς στόχους, τους οποίους θα πρέπει να εξυπηρετούν οι δαπάνες. Και εκεί θα κρίνονται κιόλας. Τα επόμενα έτη λοιπόν, σε συνεργασία με το Ελεκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς την κατεύθυνση αυτή θέλουμε να προχωρήσουμε. Κυρίε και κύριοι, ο έλεγχο του προπολογισμού περιέχει και ένα ισχυρό πολιτικό στοιχείο. Δεν είναι απλώ λογιστική η άσκηση αυτή, αλλά ε, αν τη θεωρήσουμε ενιαία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι ελεκτές του προπολογισμού, δηλαδή τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ε, φρόντισαν και πρόσεξαν πάρα πολύ να τηρηθεί εντός πλαισίων ο προϋπολογισμός και υπήρξε και μια έντονη συζήτηση για το 2013, για το διορθωτικό προϋπολογισμό και για το προϋπολογισμό του 2014 με το Συμβούλιο, ο οποίος μόλις εγκρίθηκε και αυτό είναι ένα συμβιβασμό ε, που μπορεί να μας ικανοποιεί. Ελπίζουμε ε, οι μεταφορές από χρόνο σε χρόνο να μειώνονται ε, και τα διορθωτικά και τα ταμεία συνοχής να μπορούν να χρηματοδοτούν τους αποδέκτες τους ε, λογικά χρονικά πλαίσια. Επίσης υπάρχει ένα συμβασμός μεταξύ των προτάσεων ε, του Συμβουλίου αφενός και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου Φετέρου. Και ακριβώς όταν είναι λίγοι οι πόροι, η μείωση του πολιετές δημοσιονομικού πλαισίου είναι κάτι το οποίο ε, μπορεί να υποστηριχθεί και ε, μπορεί να υποστηρίξει και τους κρατικούς προπολογισμούς. Ξέρετε, το κοινοβούλιο διαφωνεί ε, γιατί το, κατά πλειοψηφία θα επιθυμούσε αύξηση των κοινοτικών κονδυλίων. Εάν η Ευρωπαϊκή ε, ε, ε, ε, το επταετές ε, πρόγραμμα αυτό γύρω στα 900 δισεκατομμύρια είναι κάτι πολύ θετικό γιατί βλέπουμε ότι οι προϋπολογισμοί στα κράτη-μέλη αυξάνονται με δικαιολογία τον τιμάριθμο της αυξήσεις των μισθών και του κόστου ζωής, πράγμα που ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα η μείωση ε, του συνολικού προπολογισμού για το επταετές ε, πρόγραμμα σημαίνει ουσιαστική οικονομία. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ακριβώς το better spending, δηλαδή κάθε ευρώ να πιάνει τόπο, να δαπανάτε σωστά ε, και εκεί που πρέπει. Αυτά. Και έρχομαι στο τελευταίο σημείο που θέλω να αναφέρω σύντομα, 80% του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε συναρμοδιότητα, δηλαδή τα διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη και ε, οι περιφέρειες. Για την εκτέλεση λοιπόν του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρουν πολύ μεγάλη ευθύνη οι περιφέρειες και τα κράτη. Και εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τρόπο που συμμετέχουν αυτές οι αρχές. Αυτό δεν σημαίνει αντίφαση, αλλά ε, συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης. Και στο κάτω-κάτω δεν έχει σημασία από πού προέρχονται τα χρήματα, αν είναι από κοινοτικό προϋπολογισμό ε, ή εθνικό ή τοπικό περιφερειακό. Σε τελική ανάλυση είναι πάντα χρήματα των φορολογουμένων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας μερικά διαδικαστικά, σύντομα. Θα πρότεινα να υπάρχει δυνατότητα να λάβει το λόγο όποιος το ζητήσει και στο παρελθόν ε, ε, η εμπειρία ε, μας έδειξε ότι είναι καλό να δίνουμε πέντε λεπτά χρόνο σε κάθε ομιλητή για να μπορέσουν όλοι να πάρουν το λόγο και να έχουν και ένα χρόνο έτσι με ευχαίρεια να παρουσιάσουν τις απόψεις Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση για κάθε ενότητα ε, θα πρότεινα να δίνουμε το λόγο σε δύο εθνικούς βουλευτές και μετά σε έναν ευρωβουλευτή, δύο προς ένα, σε περίπτωση που το ζητήσει ο ευρωβουλευτής. Αλλά σε μια τέτοια συνεδρίαση ε, έτσι κι αλλιώς μπορούμε να δείχνουμε ευελιξία ως προς τον κατάλογο των ομιλητών. Ε, σας έχουμε δώσει κάποιες κάρτες ε, που λέγονται speaking cards και μπορείτε ε, με αυτές να ζητάτε το λόγο. Να γνωρίζουμε το όνομά σας και το κοινοβούλιο σας για να σας δίνουμε το λόγο. Αυτά νομίζω σας παρουσίασα κάπως τα πράγματα τεχνικά. Πρέπει να σας πω ότι από τις 12.30 και μετά θα ε, και ένα ε, γεύμα με σάντουιτς εδώ εκτός της αιθούσης. Θα ήθελα να δώσω το λόγο λοιπόν πρώτα στην Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού, ε, της ΕΙΜΑΣ της Λιθωανικής Βουλής. Καλώς ορίζατε θερμά, κύριε Βάικένε. Έχετε μέσα στο λόγο. Παρακαλώ. Καλημέρα σας ε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρωτοβουλία που ανέλαβε να οργανώσει αυτή την ανταλλαγή απόψεων για τα πρότυπα και, τους, και τα είδη ε, κοινοβουλευτικού ελέγχου των δημόσιων λογαριασμών. Γιατί θέλουμε να χρησιμοποιούμε με αποτελεσματικό και ορθολογικό τρόπο τα δημόσια κονδύλια και μετά την κρίση το θέμα αυτό ανέλαβε ακόμη και ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχουμε το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση το καθήκον να εξασφαλίσουμε χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και των εθνικών αλλά και των κοινοτικών κονδυλίων. Σήμερα έχω την τιμή να σας παρουσιάσω την λιθουανική εμπειρία και τα μέτρα δημοσιονομικού ελέγχου που εφαρμόζουμε στην Λιθουανική Βουλή της ΣΕΙΜΑΣ. Θα ήθελα αυτής εξ αρχής να τονίσω ότι ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των ε, δημοσίων κονδυλίων από τις αρμόδιες αρχές προβλέπονται στο καταστατικό της ε, Λιθουανικής Βουλής ε, ως πρωταρχική αρμοδιότητα της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο αποδίδουμε τεράστια σημασία σε αυτό το μέλημα του αποτελεσματικού ελέγχου των δημόσιων λογαριασμών. Στη Λιθουανία τα ευρωπαϊκά κονδύλια αλλά και οι εθνικές δαπάνες, τα εθνικά κονδύλια θεωρούνται ως κονδύλια του προϋπολογισμού. Οπότε, όταν μιλούμε για αποτελεσματική διαχείριση ε, των ε, κονδυλίων του προϋπολογισμού, εννοούμε και την ε, χρηστή διαχείριση των κοινοτικών, των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Βέβαια, έχουμε και ειδικούς επιπλέον ελέγχους για τη χρηστή διαχείριση των διαρθρωτικών κονδύλιων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίθηκαν με βάση την ενωσιακή νομοθεσία που προβλέπει ιδιαίτερες απαιτήσει σε ό,τι αφορά τον χρηστό δημοσιονομικό έλεγχο των ε, ευρωπαϊκών ενισχύσεων. Γιατί όταν μιλούμε για ευρωπαϊκά κονδύλια εννοούμε χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Γι' αυτό ακριβώς ε, και η αποτελεσματικότητα της χρήσης αυτών των κονδυλίων θα πρέπει να πληρεί ακόμη πιο αυστηρές προδιαγραφές από ότι ο, δημο, το, δημοσιονομικός έλεγχος των εθνικών δαπανών. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν τα μέτρα που ε, ε, εντάσσονται στο δικό μας δημοσιονομικό έλεγχο Έχουμε καταρχήν τον έλεγχο της απαλλαγής. Κάθε χρόνο η κυβέρνηση υποβάλλει στη Λουθανική Βουλή ένα σύνολο των ελέγχων των ε, διαφόρων εξόδων και γίνεται και δημοσιονομικός έλεγχος των συγκεκριμένων εκθέσεων καθώς και της ε, ε, νομοτυπίας των λογαριασμών. Τα αποτελέσματα αυτά στηρίζονται σε πληροφορίες που συγκεντρώνουν οι δημοσιονομικοί ελεγκτές κατά τη διάρκεια των ελέγχων και αυτές είναι η βάση για τον έλεγχο. Επίσης, οι εκθέσεις ε, των δημοσιονομικών ελεγκτών συζητώνται σε όλες τις ε, ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές. Κάθε επιτροπή ασχολείται ιδιαίτερα με τους οργανισμούς της δικής αρμοδιότητας, ενώ η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού τη Λιθωνική Βουλή εξετάζει περισσότερο οριζόντια συστημικά προβλήματα. Βέβαια, οι δικευμένε αρχέ δεν αξιοποιούν ιδιαίτερα τη διαδικασία τη απαλλαγή ω μέτρο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθολογικότητα της χρήσης ε, των ε, κονδύλιων. Δυστυχώς πολύ συχνά μιλούμε για την αρχή της ε, αποκόμισης ε, του μέγιστου αριθμού των κονδυλίων για συγκεκριμένα τομέα, ενώ η χρήση τους επαφείται στην διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης ή συγκεκριμένου Υπουργείου. Ενώ η εκτελεστική εξουσία δεν προβλέπει εναλλακτικές χρήσεις ε, για τα μη διαθέσιμα κονδύλια ή ε, για τον αντίκτυπο της μη χρησιμοποίησης τους. Θεωρούμε ότι η έλλειψη του κοινοβουλευτικού ελέγχου ουσιαστικά μετακυλεί από χρόνο σε χρόνο τα διάφορα συστημικά προβλήματα. Γιατί ξεκινούμε από απλά λογιστικά προβλήματα και, ξεκινούμε και καταλήγουμε σε συγκεκριμένες παραβιάσεις ε, του τις σχετικές νομοθεσίες και τις ε, δημόσιες προμήθειες. Θα πρέπει λοιπόν η εκτελεστική εξουσία να αναλάβει περισσότερες ευθύνες για να περιοριστεί το ποσοστό σφάλματος και η παρατυπίες ή ατασταλίες. Η η Ελέγχου του Προϋπολογισμού στις συνεδριάσεις της εξετάζει τις πιο σημαντικές εκθέσεις ε, των δημοσιονομικών ελεγκτών και έχει ακροάσει φυσικά και με εκπροσώπους των ελεγχόμενων ε, φορέων και μάλιστα διαπιστώνουμε μία μηχανή αυτών των εκπροσώπων όταν ε, καλούνται να δώσουν εξηγήσει ιδιαίτερα στην ε, κοινή γνώμη. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι αυτές οι πιέσεις είναι σημαντικές γιατί έτσι με τη λογοδοσία αυτή περιορίσαμε το ποσοστό σφάλματος των φορέων όταν καλούμε τους εκπροσώπους τους να λογοδοτήσουν, είναι πολύ πιο προσεκτικοί στον έλεγχο των λογαριασμών τους. Με την κρίση προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ. Γι' αυτό και έχουμε περιοδικούς ελέγχους συγκεκριμένων δαπανών. Ελέγχουμε ιδιαίτερα τομείς όπου θεωρούμε ότι πιο ορθολογικές και υπεύθυνες επιλογές θα μας οδηγήσουν σε οικονομίες. Οι διαχειριστές των κονδυλίων οφείλουν κάθε τρίμηνο να ενημερώνουν την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού της Λιθωνικής Βουλής για τις δαπάνες τους, για, τις, για την κατάρτιση, τις αμοιβέ των εμπειρογνωμόνων, τα έξοδα παράστασης και το καθεξής. Επίσης δίνουν λεπτομεριακές ε, πληροφορίες για τη χρήση των κονδυλίων που έχουν και τους μισθούς. Έτσι, Έχουμε ένα σύστημα ενημέρωσης με υποβολή μέσω διαδικτύου ερωτηματολογίων τα οποία χρησιμοποιούμε στη συνέχεια για να καταρτήσουμε πίνακες και να μπορούμε να αναλύσουμε καλύτερα και να συγκρίνουμε τα διάφορα δεδομένα. Η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού κάνει τις αναλύσεις και την αξιολόγηση των ε, δεδομένων αυτών. Όλα αυτά τα δεδομένα και οι αναλύσεις τους δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Λιθουανικής Βουλής. Οι θύνοντες ε, των φορέων και των θεσμικών οργάνων ε, που έχουν μεγαλύτερες δαπάνες και για τους οποίους υπάρχουν αμφιβολίες για τη χρήση τους ε, δημοσιονομική διαχείριση, καλούνται στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού για να δώσουν εξηγήσεις. Και μάλιστα πολλές φορές χρειάζεται να υποβάλουν και γραπτές αιτιολογήσεις ε, για τις δαπάνες τους. Μάλιστα έχουμε μερικές φορές και καταλόγους αποστολών για συγκεκριμένη περίοδο με τις συγκεκριμένες αμοιβέ των μελών των αντιπροσωπιών και με αιτιολόγηση της ανάγκης πραγματοποίησης συγκεκριμένης αποστολής ή επίσκεψης. Επίσης κάνουμε αναλύση των δαπανών και των αμοιβών ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Θέλουμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια το κόστος των υπηρεσιών αλλά και την προστιθέμενη αξία και τη χρησιμότητά τους. Και μάλιστα για τους φορείς που οι αναλύσεις ε, των δαπανών έγιναν με πολύ διεξοδικό τρόπο, ε, διαπιστώσαμε μία δυσαρέσκεια γιατί οι εκπρόσωποι τους ε, έδωσαν λόγο όχι μόνο στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού αλλά λογοδότησαν και δημοσίως. Παρ' όλα αυτά όμως διαπιστώσαμε ότι στη συνέχεια οι δαπάνες τους μειώθηκαν γιατί χρειάστηκε να δώσουν πιο λεπτομεριακές εξηγήσεις για την αιτιολόγηση αυτών των δαπανών. Σε ό,τι αφορά την εξέταση των μισθών, εκεί δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις, ε, στους δημοσιονομικούς κανόνες, ιδιαίτερα για, για τα επιδόματα. Γιατί με την κρίση είχαμε μία μείωση μισθών και περικοπές επιδομάτων. Θα πρέπει βέβαια ταυτόχρονα να δώσουμε κίνητρα στους εργαζομένους και μερικές φορές τα επιδόματα είναι ένα επιπλέον κίνητρο. Αλλά πολλές φορές η χορήγηση των επιδομάτων υπακούει σε υποκειμενικά κριτήρια. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι σε χαλεπούς καιρούς ε, δημοσιονομικής κρίσης η θέσπιση αυτών των επιδομάτων και των, πριμ, των είναι αδικαιολόγητη και απαράδεκτη. Και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη σε κάθε εξέταση προϋπολογισμού. Για παράδειγμα, πέρυσι διαπιστώσαμε ότι ένα πανεπιστήμιο κατέβαλε 3,5 εκατομμύρια του Εθνικού μας Νομίσματος σε τέτοιες πρημοδοτήσεις και εμείς ε, για την επόμενη χρονιά μειώσαμε την χρηματοδότηση αυτού του ε, πανεπιστημίου κατά 3,5 εκατομμύρια. Γιατί θεωρούμε ότι σε περίοδο κρίσης δεν επιτρέπονται τόσο παχυλές ε, πρημοδοτήσεις. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνεται μια πιο ορθολογική χρήση των κονδυλίων. Τέτοιου είδου κίνητρα όπω τα επιδόματα και οι πρημοδοτήσει θα πρέπει σε περίοδου κρίση να περικόπτονται οι οικονομίες αυτές ε, ήδη έχουν αποφέρει καρπούς, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η κοινή γνώμη περιμένει με αδημονία τέτοιου είδους ε, εξηγήσει και εκθέσεις. Και μερικές φορές ε, δακτυλοδεικνύονται οι υπερβολικά σπάταλοι ηθήνοντες και καλούνται να λογοδοτήσουν και δημοσίως. Θα πρέπει τα διάφορα θεσμικά όργανα και οι δημόσιοι φορείς να είναι υπόλογοι στους πολίτες. Έχουμε και το ανώτατο ελεκτικό φορέα και το έργο του συμβάλλει στην ε, πιο ορθολογική και χρηστή διαχείριση των κονδύλιων. Όλοι αυτοί οι δημοσιονομικοί έλεγχοι αναλύουν και τις αποδόσεις ε, των διαφόρων συστημάτων. Οπότε, σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελαττώματα στη λειτουργία του συστήματος, ή τα ελαττώματα αυτά διορθώνονται και έτσι εξασφαλίζεται πιο αποτελεσματική διαχείριση των κονδυλίων. Με τους δημοσιονομικούς αυτούς ελέγχους εξετάζουμε και την ορθολογικότητα συγκεκριμένων δαπανών. Γιατί το καταστατικό εσωτερικό κανονισμό τη Βουλή χορηγεί στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού την αρμοδιότητα ελέγχου όλων αυτών των ε, εκθέσεων των δημοσιονομικών ελεκτών. Και όταν έχουμε εκθέσεις και για την απόδοση, τις στέλνουμε στην αρμόδια καθήλυνη επιτροπή. Εκείνη εγκύπτει στο θέμα της λειτουργίας του συστήματος, ενώ η δική μας Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ασχολείται με την αποτελεσματικότητα της χρήσης των διαφόρων κονδυλίων. Γιατί διαπιστώνουμε ότι οι δικευμένες επιτροπές, οι κοινοβουλευτικέ επιτροπές, δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την πτυχή αυτή. Μετά την ε, έκθεση, τις εκθέσεις λοιπόν των δημοσιονομικών ελεκτών και μετά από ακροάσεις των εκπροσώπων των διαφόρων φορέων για να δούμε κατά πόσο ακολουθούν τις συστάσεις η Επιτροπή μας εκφράζει την πολιτική στήριξη προς τις συστάσεις και ζητά και ενημέρωση και τακτικές εκθέσεις για την εφαρμογή των συστάσεων. Έτσι ασκείται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ του ελεγχόμενου φορέα και του ελεγκτικού φορέα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή κάποιων συστάσεων, το Κοινοβούλιο δίνεται να εγκρίνει ψήφισμα που θα έχει δεσμευτικό και υποχρεωτικό χαρακτήρα. Η εφαρμογή αυτού του ψηφίσματος ελέγχεται από το ίδιο το Κοινοβούλιο. Μερικές φορές τέτοια ψηφίσματα είναι το μοναδικό μέσο για να εξασφαλίσουμε συμμόρφωση με τις συστάσεις ε, του δημοσιονομικού ελέγχου. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών προβλέπει και κάποια κονδύλια για τις κρατικές επενδύσεις. Πρόκειται για κονδύλια που χρησιμοποιούνται για έργα υποδομών, για δημόσιες προμήθειες και για εξυγχρονισμό του των μέσων πληροφορικής. Ενώ η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού ασκεί την εποπτεία στην εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων. Επίσης, η Επιτροπή μας ενδιαφέρεται ε, για την ε, επιτόπη ε, εφαρμογή αυτών των σχεδίων. Γι' αυτό και πραγματοποιούμε ελέγχους επιτόπου για να εξασφαλίσουμε την χρηστή διαχείριση στη χρήση αυτών των κονδύλιων. Μετά από ανάλυση της κατάστασης, η Επιτροπή μας εκπονεί ε, σχέδιο απόφασης με προτάσεις και συστάσεις προς τις αρμόδιες αρχές. Επίσης, ε, η Επιτροπή μας ε, έχει διακριτική ευχαίρεια ως την επιλογή των ελεγχόμενων προγραμμάτων. Η επιλογή αυτή γίνεται με βάση πληροφορίε που λαμβάνουμε από διάφορες πηγές και κυρίω καταγγελίε για πιθανή αναποτελεσματικότητα ή παρατυπία στη χρήση των κονδύλιων. Και τώρα να σας παρουσιάσω τον τρόπο ελέγχου των διαρθρωτικών κονδύλιων και να σας ε, δώσω με περισσότερες λεπτομέρειες για τις αρμοδιότητες των ελεκτικών φορέων. Το 2006, όταν εκπονήσαμε αυτό το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των διαρθρωτικών ε, κονδυλίων και ενισχύσεων αποφασίσαμε να αναθέσουμε στον ανώτατο ελεκτικό φορέα της Λιθουανίας την αρμοδιότητα του δημοσιονομικού ελεγκτή και για τα διαρθρωτικά κονδύλια. Από ό,τι ξέρω, μόνο η Ρουμανία έχει εφαρμόσει ένα αντίστοιχο μοντέλο. Οι άλλες χώρες μέλη έχουν αναθέσει σε άλλους οργανισμούς και φορείς αυτή τη λειτουργία. Η Λιθουανία όμως διάλεξε το συγκεκριμένο μοντέλο για πολλούς και διάφορους λόγους. Το μοντέλο δηλαδή της ΕΠΑ της αρχής. Καταρχήν, ο φορές αυτός, ο υπατός ελεκτικός φορές, είναι ανεξάρτητος σε σχέση με τους άλλους ελεκτικούς φορείς. Η ανεξαρτησία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ε, αποτελεσματική εκτέλεση του έργου. Επίσης, ε, η Λιθουανία λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ανάγκη χρηστής διαχείρισης ιδιαίτερα των διαρθρωτικών κονδύλιων. Γι' αυτό και διαλέξαμε μία διάρθρωση ε, για την οποία δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του φορέα. Θέλουμε επίσης να καθησυχάσουμε και την πολιτική μας τάξη αλλά και την κοινή γνώμη και να αποφύγουμε διαρθρωτικά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη χρήση των κονδύλιων. Και μάλιστα μπορούμε ήδη να διαπιστώσουμε, αν βασιστούμε στην εμπειρία μας, ότι αυτό το ανώτατο ελεγκτικό όργανο ολοκλήρωσε την εργασία του πολύ ε, ενδελεχώς και εξαιρετικά αυστηρά. Έχει εντοπίσει τα διευθυντικά προβλήματα και απέτησε να καταργηθούν. Και ακριβώς λόγω αυτής της μεγάλης ευσυνειδησίας αλλά και της αργής αντίδρασης από πλευράς των άλλων θεσμών για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, Λόγω όλων αυτών λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακύρωσε, ανέστηλε μάλλον το 2011 την καταβολή ενός τμήματος των ενισχύσεων προς τη Λιθουανία, πράγμα που προκάλεσε σημαντικό σκάνδαλο. Τελικά όμως ε, ήταν θετικός αντίκτυπος για την κατάσταση διότι έτσι λήφθησαν οι απαραίτητες αποφάσεις ώστε να τελειοποιηθεί το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και το 2012 αυτό το θεσμικό ελεγκτικό όργανο όργανο τελικά ε, παρουσίασε, μπόρεσε να παρουσιάσει θετική ε, κατάσταση πια. Δεδομένου ότι το 2012-2013 οι δηλωμένες δαπάνες έφτασαν στο ψηλότερο επίπεδο, θεωρούμε ότι χάρη στον νότο το ελεκτικό μας όργανο η κατάσταση βελτιώθηκε και ο θεσμός αυτός συνέβαλε ώστε η Λιθουανία να μην έχει προβλήματα λόγω ε, κακής λειτουργίας του συστήματος ή λόγω των, της δήλωσης δαπαν, μη επιλέξιμων δαπανών. Ίσως να υπάρχει κόσμος που να θεωρεί που ένας θεσμός που είναι θεωρητικά ανεξάρτητος ε, ε, είναι λιγότερο αυστηρός, μπορεί να μην παρατηρήσει τις μικρές ε, τα μικρά λαθάκια θα ήταν καλύτερα γιατί αυτό θα είχε μπορέσει να μας, ε, ε, να μας γλιτώσει από τις δυσάρεστες εξηγήσεις μπροστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ πιστεύω ωστόσο πως η επιλογή ήταν δύσκολη, μας δημιούργησε προβλήματα αλλά μας κατέστησε δυνατότερους και γι' αυτό και επιλέξαμε το ίδιο μοντέλο για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και επίσης επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εμπιστοσύνη στο ελεγκτικό μας αυτό όργανο δεν παρουσίασε παρατηρήσεις και ανέκαθεν ενέκρινε την ετήσια έκθεση αυτού του θεσμικού οργάνου. Μπορούμε λοιπόν να ελπίζουμε πως Κατά τη διάρκεια της περίοδου 2014-2020 ο έλεγχος της χρήσης των διευθυντικών ταμείων θα είναι σωστός πια. Θα να προσθέσω ότι οι ετήσιες εκθέσεις εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εκθέσεις αυτές συζητώνται στο πλαίσιο της ε, Ελεγκτικής Επιτροπής ε, του Κοινοβουλίου. Ε, η Επιτροπή μας κάνει ό,τι μπορεί ώστε οι συστάσεις που παρουσιάζονται από τους ελεγκτές να εφαρμόζονται εγκαίρως. Χαιρόμαστε που η Λιθουανία έχει τώρα ένα σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που επιτρέπει την εξασφάλιση της υπεύθυνης χρήσης των κοινωτικών κονδυλίων. Εν τέλει, να σας θυμίσω πως η Ελεγκτική Επιτροπή του ε, Λιθανικού Κοινοβουλίου προβαίνει και μάλλον ε, κάνει ένα μεγάλο έργο ελέγχου των δαπανών και χρησιμοποιεί ένα σωρό μέσα, έλεγχος της εκτέλεσης του προπολογισμού, έλεγχος της έκθεσης ελέγχου, ε, λογιστικού ελέγχου, έλεγχος της έκθεσης απόδοσης, εξασφαλίζουμε την εποπτεία και την εφαρμογή, προβαίνουμε στην παρακολούθηση των ε, επισφαλών δαπανών και επίσης η Επιτροπή αυτή έχει ορίσει και το ανώτατο θεσμικό όργανο οικονομικού και λογιστικού ελέγχου ε, που με τη σειρά του προβαίνει στην ανάλυση των εκθέσεων που παρουσιάζει το όργανο αυτό. Να σημειώσουμε επίσης ότι για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων έχουμε όχι μόνο ένα εργαλείο ε, αυτό το εργαλείο, αλλά και βασιζόμαστε και στην διαφάνεια. Να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Εύχομαι καρποφόρες εργασίες, ε, εύχομαι να προκύψουν νέες ιδέες και όλα αυτά έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον κεντρικό μας στόχο, δηλαδή την ε, λογική, ορθολογική και αποτελεσματική χρήση των δημοσιονομικών πόρων, καθώς επίσης την ενίσχυση της ευθύνης της εκτελεστικής εξουσίας στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βάικενε για αυτές τις ενδιαφέρουσες απόψεις και την παρουσίαση της εργασίας ε, της Επιτροπής σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης και τη μεγάλη ειλικρίνεια με την οποία παρουσιάσατε ε, τις διαδικασίες βελτίωσης μετά από κάποιες δυσκολίες που είχαν διαπιστωθεί. Νομίζω είναι ένα πάρα πολύ εύγλωτο παράδειγμα και είμαστε εδώ για να διδασκόμεθα κι ένας από τον άλλον και να μιμούμαστε το καλό παράδειγμα. Θα ήθελα να σας πω ότι έχετε μια πράσινη σελίδα που είναι ένα έντυπο και μπορείτε να το συμπληρώνετε για να σας δίνουμε το λόγο. Λέγεται Speaking Note ε, και παρακαλώ να τους συμπληρώσετε αν θέλετε να ζητήσετε το λόγο. Λοιπόν, θα δώσω πρώτα το λόγο από Εθνικό Κοινοβούλιο τώρα ε, στον κύριο Γκρούτκοβιτς από την Κροατία. Παρακαλώ, δεν σας βλέπω κιόλα Πού κάθεστε. Ε? Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους. Ε, έρχομαι από την ε, Κροατική Βουλή και θα ήθελα να σας αναφέρω και τις δικές μας εμπειρίες στο δημοσιονομικό ελέγχο. Γιατί όπως είπαμε, ο δημοσιονομικός ε, έλεγχος είναι πολύ σημαντικός, όχι μόνο τώρα λόγω της ύφεση, αλλά είναι σημαντικό το θέμα της λογοδοσίας των πολιτικών απέναντι στους πολίτες. Ένα από τα θεμελιώδη σημεία που έχουμε και κάνουμε αυτή τη στιγμή στην Κροατία είναι ότι το κρατικό γραφείο ε, που είναι για τον έλεγχο που είναι αρμόδιο για την ε, νομοτυπία και την αποτελεσματικότητα των ε, κονδυλίων και των εθνικών και των τοπικών φορέων. Αυτό το κάνει για τα προηγούμενα χρόνια και μετά την ανάλυση των προηγούμενων χρόνων και των δαπανών των προηγούμενων χρόνων και μετά την ε, είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσαμε ε, όταν γίνεται ο έλεγχος ε, των φορέων να υποβάλλεται στην Κρατική Βουλή και στην αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού της Κρατικής Βουλής η έκθεση με τον απολογισμό όλων των ελεγχόμενων φορέων. Έτσι γνωρίζουμε τι κάνει αυτό το ελεκτικό συνέδριο της Κροατίας ή ο ελεκτικός φορέας. Και η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή είναι ε, η Επιτροπή των Οικονομικών. Δεν έχουμε ειδική επιτροπή ελέγχου του προϋπολογισμού στην Κρατική Βουλή. Και όπως είπε και η εκπρόσωπος από τη Λιθουανία, και το δικό μας κοινοβούλιο μπορεί να επαναφέρει στην τάξη καλώντας να λογοδοτήσουν τους εκπροσώπους των ελεγχόμενων φορέων. Και αυτό συνιστά σημαντική βελτίωση γιατί μέχρι στιγμής ο θεσμικός φορέας που ασχολείται με τους ελέγχους απλώς ενημέρωνε την κρατική βουλή για το έργο του. Μερικές φορές όμως αυτή η ενημέρωση γινόταν ε, κάπως καθυστερημένα. Μπορούσε να καθυστερήσει και έναν ολόκληρο χρόνο δεν ήταν επίκαιρη δηλαδή. Τώρα με το που ολοκληρώνεται ο έλεγχος ενός θεσμικού οργάνου, η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Οικονομικά και τον Προϋπολογισμό συνέρχεται και εξετάζει αμέσως την έκθεση ώστε να ζητήσει διόρθωση των ατασταλιών. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο και για το δημοσιονομικό έλεγχο, για τον έλεγχο του προϋπολογισμού για την τρέχουσα πια διαχειριστική χρήση και όχι για τις προηγούμενες. Και αυτό γίνεται ύστερα από καταγγελία, είτε από θεσμικό φορέα, είτε από πολίτη. Έτσι, ελέγχουμε την κατάσταση πια για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση. Έχουμε λοιπόν από τη μια το Υπουργείο Οικονομικών που πραγματοποιεί δημοσιονομικό έλεγχο και αφετέρου έναν ανεξάρτητο φορέα που είναι το Εθνικό Γραφείο Ελέγχου που ασκεί το δημοσιονομικό έλεγχο. Έχουμε λοιπόν έναν αποτελεσματικό έλεγχο του προϋπολογισμού μας. Γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός μας ρόλος. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ πολύ ε, το πρόεδρο ε, της αρμόδιας κρατικής επιτροπής για τον έλεγχο του προπολογισμού και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο ε, σε κάποιον από το Ρίξτακ, το Σουηδική Βουλή, που είναι ο κύριος Γιώνας Γιάκομψεν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, ζήσαμε μια μεγάλη οικονομική κρίση στις αρχές της δεκαετίας του 90 εμείς. Και η τωρινή παγκόσμια κρίση που ήρθε αργότερα, εμάς μας είχε επισκεφθεί πριν από 18 χρόνια. Και οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ε, ο τομέας των ακινήτων είχαν πληγεί ε, βαθύτατα από την αρχή της δεκαετίας του 90 με κάποιες κατασκευαστικές ε, στεγαστικές εταιρείες οι οποίες επτόχευσαν από τη μια μέρα στην άλλη και χρειάστηκε μαζική επέμβαση της κυβέρνησης για να κεφαλαιοποίηση των τραπεζών πράγμα που είχε ελεύθερα αποτελέσματα στα οικονομικά μας. Έκτοτε λοιπόν έβημεν σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων. Μεταρρυθμίσαμε όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις τράπεζες και το χρηματοπιστωτικό τομέα αλλά και το δημόσιο ε, για να μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα όλη αυτή τη διαδικασία και τη δημοσιονομική. Θα ήθελα να πω επίσης ότι θελήσαμε να διατηρήσουμε στα χέρια του Κοινοβουλίου ένα στοιχειώδη έλεγχο ε, των ε, δημοσίων δαπανών. Ε, αυτό είναι χρηστή οικονομική διαχείριση. Να έχουμε λόγο όχι μόνο εκ των υστέρων για τον έλεγχο του προπολογισμού, αλλά και στην κατάρτιση του προπολογισμού εκ των προτέρων. Ε, θα πρέπει πάντα να έχει στα χέρια του το κοινοβούλιο τον έλεγχο του προπολογισμού σε όλα τα στάδια. Αυτό λοιπόν που επιλέξαμε να ε, πράξουμε ήταν να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη επιρροή στην κατάρτιση του προπολογισμού και να μην αφήνουμε ε, μεγάλη ελευθερία στην κυβέρνηση. Και εκ των υστέρων έλεγχος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού είναι σημαντικός, αλλά για μας σημαντικότερο είναι το πρώτο στάδιο. Έχουμε λοιπόν μία προσέγγιση σε δύο χρόνους, σε δύο φάσεις. Αυτή η πρακτική έχει τώρα κατοχυρωθεί και με νομοθεσία και βελτιωθεί και τελειοποιηθεί, αν θέλετε, την τελευταία 20 αιτία. Το 2008-2009 εξέσπασε η επόμενη νέα χρηματοοικονομική κρίση. Εμείς συνεχίσαμε τις μεταρρυθμίσεις και πιο πρόσφατα ε, υιοθετήσαμε μια νέα μεταρρύθμιση με τα εξή στοιχεία. Πρώτον, προσπαθούμε να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, κυρίως στο δημόσιο τομέα, και ε, η κυβέρνηση έχει θέσει και στόχους για ε, οικονομίες στις δαπάνες της. Η ε, Σουηδική Βουλή διατήρησε αυτό το στόχο, 1% του ΟΕΠ κατά μέσο όρο ανά κύκλο της ε, οικονομικής συγκυρίας. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι το κράτος μπορεί κάλλιστα να έχει ένα χρόνο έλλειμμα υπό την προϋπόθεση ότι την επόμενη χρονιά θα το ίσως και λύσει και θα το υπερσκελίσει μάλιστα κατά 1% μια ποσοστιαία μονάδα του προϋπολογισμού για να μπορεί στη συνέχεια να το κατανείμει στις δαπάνες. Στο ε, ε, οικονομικό νόμο για τον προϋπολογισμό Επίσης ε, είχε αποφασιστεί από τη Βουλή να μπει μια οροφή στις συντάξεις ε, μέσα σε μια τριετία. Υπάρχει λοιπόν ένα πλαίσιο δαπανών, φορολογίας, ε, προγραμματισμένου πλεονάσματος στον προϋπολογισμό και η κυβέρνηση έχει κάποια δυνατότητα και διακριτική ευχαίρεια να δράσει. Τα ίδια ισχύουν και για την τοπική αυτοδιοίκηση και τις περιφέρειες. Από το 2000 είναι υποχρεωμένοι να έχουν ισοσκελισμένο προπολογισμό. Σε περίπτωση ελλείμματος, στην επόμενη τριετία μέσα πρέπει αυτό να έχει λυθεί. Είναι λοιπόν αρκετά σφιχτές αυτές οι δημοσιονομικές διαδικασίες. Και συγκεκριμένα στις Σεπτεμβρίου, το αργότερο, θα πρέπει να κατατίθεται στη Βουλή ε, το σχέδιο προϋπολογισμού. Ακολουθεί μελέτη αυτού σε δύο φάσεις. Πρώτα το γενικό πλαίσιο, το γενικό προσανατολισμό ε, και μάλιστα ε, σε 20 κατηγορίες εξετάζουμε τα έσοδα και τις δαπάνες κατανεμημένες με πάντα μία οροφή, ένα ανώτατο όριο. Αυτό λοιπόν γίνεται σε μία φάση ενιαία και το πλαίσιο και οι δαπάνες ορίζονται από το Κοινοβούλιο για 20 διαφορετικές κατηγορίες. Έτσι λοιπόν έχει το γενικό πλαίσιο. Στη συνέχεια ασχολούμαστε με τις διάφορες θέσεις του πυροπολογισμού, Το κάθε κονδύλι χωριστά το εξετάζουμε λεπτομερώς. Τι σημαίνει αυτό. Όταν έχουμε αύξηση σε μία πίστοση του προϋπολογισμού ε, θα πρέπει στην ίδια κατηγορία αυτή να συνοδεύεται και να αντισταθμίζεται από αντίστοιχη μείωση κάπου αλλού. Στο παρελθόν αυτό δεν γινόταν. Και μέχρι τα Χριστούγεννα το αργότερο θα έχει τελειώσει η εξέταση του προϋπολογισμού κάθε φορά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί έτσι ελέγχουμε τις δαπάνες πάντα πριν ε, από την εκτέλεση του προϋπολογισμού, στην κατάρτισή του. Το δεύτερο στοιχείο είναι τώρα η παρακολούθηση της εκτέλεσης. Ωραία, εγκρίναμε αυτά τα κονδύλια, πώς ε, δαπανώνται αυτά. Γίνεται αυτός ο έλεγχος σε εθνικό επίπεδο πάντα ε, υπό τον έλεγχο του Κοινοβουλίου, αλλά από ανεξάρτητη μονάδα, από ανεξάρτητη υπηρεσία με οικονομικό έλεγχο και μάλιστα είναι διτός αυτός. Ε, ελέγχουν όλο το κράτος, την κυβέρνηση, την κεντρική, την κεντρική τράπεζα, και τα λοιπά. Και το, δεύτερο ε, σκέλος είναι όχι ο αμυγής οικονομικός έλεγχος, αλλά ο έλεγχος αποτελεσματικότητας. Δηλαδή, επιλέγουμε κάποιους τομείς και κοιτάμε πιο λεπτομέρως, όχι εμείς, η αρμόδια αρχή, ε, ε, με ποιο τρόπο εκτελείται ο προπολογισμό και αν είναι πραγματικά εύστοχες οι δαπάνες και αν έχει ε, πιάσει τόπο η κάθε κορώνα που έχει δαπανηθεί. Όλα αυτά υπό την γενική αιγίδα και τον έλεγχο του Κοινοβουλίου τελικά. Συνοψίζω. Συμμετέχουμε στην κατάρτιση του προϋπολογισμού αλλά και ε, στον έλεγχο της ε, ελέγχουσας αρχής της οικονομικής επιθεώρησης ας πούμε. Και έτσι ελέγχουμε πάρα πολύ καλά και την οικονομία και τις δαπάνες. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση της κατάστασης στη Σουηδία και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλω να δώσω το λόγο στη συνάδελφο την κυρία Ινγκέ Γκρέσλερ. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους που μίλησαν. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Θα ήθελα να πω από πλευρά του εισηγητού γιατί σκεφτήκαμε αυτή τη συνάντηση και πώς θέλουμε και πρέπει να εντείνουμε τη συνεργασία μας. Το Σεπτέμβριο του 2012 για πρώτη φορά λάβαμε ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία ε, του κοινοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2012. Αυτό το καλωσορίζουμε ρητά, αγωνιστήκαμε άλλωστε γι' αυτό. Και τι μας λέγουν αυτοί οι αριθμοί, ότι το 2012 οι πληρωμές ήταν 140 δισεκατομμύρια περίπου και για 4,419 δισεκατομμύρια χρειάστηκαν οικονομικές διορθώσεις. Και από αυτά η πραγματική ανάκτηση ήταν 678 εκατομμύρια ή 3,2% των πληρωμών. Γύρισα πίσω σε ζεστό χρήμα δηλαδή από τις απαιτήσει που είχαμε. Εδώ χρειαζόμαστε τα εθνικά κοινοβούλια. Γιατί τελικά ο εθνικός φορολογούμενος πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη όταν υπάρχει πρόβλημα στα ε, ενωσιακά οικονομικά. Το 58% όλων των ε, διορθώσεων αφορούν μία χώρα, ε, την Ισπανία για την περίοδο 2000-2006, την προγραμματική. Τρία ήταν τα κράτη-μέλη που οφείλονται για, ε, οφείλονται 80% των ασφαλμάτων ε, στην περιφερειακή πολιτική και είναι με τη σειρά οι χώρες Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα. Και στην επόμενη περίοδο 2006-2013 έχουμε αυτές τις τρεις ηγετικές χώρες εντός εισαγωγικών όπου η Ελλάδα πλέον έχει ξεπεραστεί από την Τσεχία, Πολωνία και Ρουμανία. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό, μήπως δεν γίνονται έλεγχοι ε, τόσο καλοί στην Ελλάδα ή μήπως έχουν επιδεινωθεί άλλες χώρες για να την ξεπεράσουν, δεν ξέρω, θα το βρούμε. Ε, τι θέλουμε να πούμε εμείς με τους αριθμούς, ότι λίγες είναι εκείνες οι χώρες που έχουν μεγάλα λάθη και σφάλματα ε, στα διαρθρωτικά και στη συνοχή και δυσκολεύουν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς επειδή είναι υπεύθυνε πολύ λίγες χώρες για πολύ μεγάλα σφάλματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι κάνει ως αντίδραση. Καλεί όλους να βελτιώνουν τα συστήματά τους. Το 80% του προϋπολογισμού της Ένωσης όμως είναι στη συνδιαχείριση. Είναι συντρέχουσα αρμοδιότητα και θα μας πει και το ελεκτικό συνέδριο στη συνέχεια ότι κάθε χρόνο βλέπουμε ότι το 60% θα μπορούσε να είχε αποφευθεί αυτό το λαθόν αν λειτουργούσαν σωστά τα συστήματα των κρατών μελών. Γι' αυτό βλέπουμε ποιο είναι το κοινό μας έργο. Πώς θα κάνετε εσείς τις δικές σας κρατικές αρχές να λειτουργούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά έτσι ώστε η έλεγχη να είναι σωστή. Να μην έχουμε αυτή τη στρεβλή εξέλιξη. Όλοι διαμαρτύρονται για τους βαρύς ε, ε, ευρωπαϊκούς ελέγχους, ότι είναι πολύ συχνή και πολύ επώδυνοι, αλλά τι κάνουμε για να το αποφύγουμε αυτό. Ε, καλέσαμε τον αρμόδιο Ισπανό Υπουργό στην Επιτροπή μας και είχαμε και συνομιλίες με τους ομολόγους του από την Τσεχία και τη Ρουμανία διοργανώσει. Χάρη στον συνάδελφο Γκάιερ που το είχε κάνει και πέρσι αυτό τα κράτη-μέλη τίθενται πρώτον ευθυνών τους, αυτό είναι το ένα. Αλλά μετά από 20 χρόνια εσφαλμένων υπολογισμών κάτι πρέπει να κάνει περισσότερο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μεγαλύτερη συνέπεια από ό,τι στο παρελθόν. Η Ισπανία 19 χρόνια πλέον είναι στην κορυφή και μαζί με την Ιταλία των λαθών και των σφαλμάτων. Μα καλά είμαστε και κορόιδα αλλά υπομονητικά κορόιδα. Η, ε, Ο ε, κανονισμός ε, των ε, διαρθωτικών ταμείων επιτρέπει όταν υπάρχει ένα πρόβλημα να διορθώνεται από κάποια άλλη κατηγορία. Αλλά ουσιαστικές συνέπειες δεν υπάρχουν. Όταν γίνονται λάθη στην περιφερειακή στήριξη παραμένουν τα πάντα όπως έχουν. Αν το συγκρίνουμε με κάποιες κυκλοφοριακές παραβάσεις, ε, αν κάναμε ό,τι κάνουμε στην οδική κυκλοφορία, μερικές χώρες δεν θα είχαν δικαίωμα να οδηγούν καν, θα τους είχαμε πάρει το δίπλωμα με βάση το point system και τις ε, ε, ποινές και τα πρόστιμα που επιβάλλονται και οι χώρες που δαπανούν σωστά πληρώνουν, καταβάλουν στον γενωτικό προπολογισμό, συνεισφέρουν ε, και μετά καλούνται να διορθώσουν και τα στρεβλά των κρατών που κάνουν λάθη. Ελπίζω να είναι κάποιος παρόν από την Ιταλία, γιατί είναι σπεσιαλίστη η Ιταλία σε αυτά τα θέματα. Είδαμε ένα έργο με 300 εκατομμύρια ε, λάθη που έγιναν, τα οποία επιβάρυναν τον ε, Ιταλικό κρατικό προϋπολογισμό. Δεν ε, επιβαρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν βοηθάει κανένα να υπάρχει τέτοια διασπάθηση και τέτοια κακοδιαχείριση, ούτε στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Χρειάζεται ένας αυτοματισμός για καθαρές διορθώσεις των δημοσιονομικών και ε, οι χώρες που έχουν υψηλά σφάλματα θα πρέπει να πιεστούν να γίνουν αυτά. Τώρα το επιτρέπει ε, ο κανονισμός και θα πιέσουμε πάρα πολύ να μειωθεί το ποσοστό των σφαλμάτων. Θέλουμε μία διαδικασία όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάλογα με το ποσοστό σφάλματος να αναπτύσσει και να κάνει ιδιαίτερους ελέγχους για ε, την ελόγω χώρα. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άμεσα να τα ελέγχει αυτά. Εάν διαπιστώνει λοιπόν η Κομισιόν ότι ακόμα και αν τα έργα που έχουν ε, πιστοποιηθεί από τις χώρες, δηλαδή έχουν εγκριθεί, ελεγχθεί και θεωρούν ότι είναι ελεύθερα ασφαλμάτων, θα πρέπει να ελέγχεται και με καταποκοπή μειώσεις, αυτό πάνω από 3%, γιατί μόνο 3% υποχρεούνται να επιστρέφουν τα κράτη δεν είναι αποτελεσματικό, γιατί θα τους πονέσει περισσότερο αν είναι αναλογικό του σφάλματος το ποσοστό και να μην έχει μια όροφη 3%. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη λοιπόν που δεν εφαρμόζουν σωστά ε, τον κοινοτικό προπολογισμό και αυτό διακυβεύει την αποτελεσματικότητα του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μας είναι σημαντικό αυτό το θέμα και ελπίζουμε να υπάρχει μια κοινή συνεργασία σας. Ευχαριστώ πολύ. Ja, vielen Dank, äh, Frau Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρέσλε. Είναι συντονίστρια στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και ανέφερε μερικά ζητήματα που μας απασχολούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μας ανησυχούν, αλλά και μας δυσκολεύουν. Πρόκειται και για αρμοδιότητες τώρα των κρατών μελών. Και θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων που θέλουν να πάρουν από αυτού το λόγο. Χρόνο έχουμε ακόμα σε αυτή την πρώτη συζήτηση και να καλωσορίσω εδώ τον Πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου, τον κύριο Καλτέρα. Καλωσορίσατε τη συνεδρίασή μας. Τότε να δώσω το λόγο σε κάποιον εκπρόσωπο ε, της, ε, της Βουλής ε, της Ιταλίας, τον κύριο Φραντσέσκο Καριέλο. buongiorno a tutti. Καλημέρα σε όλους. Εγώ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, συνάδελφοι, κάποιες σκέψεις όσον αφορά το πρόβλημα που, ε, που έχει ε, προκύψει, γιατί νομίζω ότι δημιουργείται πριν από τα πριν φτάσει στα κοινοβούλια, δηλαδή ε, το έλεγχο των δημοσίων δαπανών και την απόκληση ανάμεσα στις δικές μας αποφάσεις ως νομοθετών και των ε, τεχνικών οργάνων που είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο. Πολύ συχνά η οικονομική διαχείριση έχει δεχτεί επικρίσεις ε, και δικαίως για ε, έλλειμμα δημοκρατικό λόγω των αποφάσεων που λαμβάνονται σε εθνικό, στο ευρωπαϊκό επίπεδο και το, σχέση τους με το εθνικό επίπεδο. Αυτή η προσοχή δίνεται και στις, ε, μάλλον αυτό, αυτή η κατάσταση επηρεάζει και τις σχέσεις ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και τους άλλους εθνικούς θεσμούς. Υπάρχουν βέβαια θέματα που είναι καθαρά τεχνικά και αυτά ανατίθεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένα και ανεξάρτητα όργανα. Στη δική μας περίπτωση πρόκειται για την Ίστατ που είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής το οποίο παρέχει τα στοιχεία στην Eurostat και άρα και στην Κομισιόν για τους στόχους της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας. Αντιθέτως δεν είναι αποδεκτό η Εθνική ε, Τράπεζα ή τα Υπουργεία ή τα τεχνικά τους τμήματα επικαλούμενα την ευρωπαϊκή πειθαρχία να δίνουν, μάλλον να αποκλείουν, μάλλον να αναλαμβάνουν αρμοδιότητες που έχουν μόνο οι νομοθέτες. Η τα τεχνικα του τμηματα επικαλουμενα την ευρωπαικη πειθαρχια να δινουν μαλλον να αποκλειουν δηλαδή τα όσα προβλέπονται στο Fiscal Compact και στο εξαπλό πακέτο ε, μέτρων ε, ε, οδηγούν στη δημιουργία του οργανισμού για τον έλεγχο της οικονομίας. Όπως ξέρετε η Ιταλία έχει μείνει λίγο πίσω σε αυτήν την εξέλιξη. Ήταν τελευταία χώρα που ευθυγραμμίστηκε και ίσως να πληρώνουμε αυτή την καθυστέρηση. όσον αφορά την έλεγχο και την επαλήθευση των εθνικών μας λογαριασμών. Όλα αυτά λοιπόν ε, έγιναν τώρα. Εντός λίγο θα γίνει η ψηφοφορία και έχει περάσει από τα δύο σώματα ώστε να μας συμβουλεύσουν οι βουλευτές μας που είναι ειδικοί για την δημόσια οικονομία. Ελπίζουμε λοιπόν ότι με τη δημιουργία αυτού του οργάνου οι ελεκτικές μας δυνατότητες για τους ελέγχους, αλλά και για, έλεγχους αλλά και για την δημόσια οικονομία ε, θα είναι πιο αποτελεσματική. Μέσω λοιπόν αυτής της νομοθεσίας που εγκρίθηκε το 2012 η υπηρεσία μας ε, δεν, έχει ακόμα, ε, δεν λειτουργεί ακόμα και αυτό λόγω ορισμένων τεχνικών ε, υπουργικών δομών που με πράγματα τα οποία γίνονταν από την Εθνική μας Τράπεζα αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών και που έχουν παίξει στην ουσία το ρόλο των ε, αξιολογητών και πρόκειται εδώ για μια προφανή ε, σύγκρουση ανάμεσα στη τεχνική και την πολιτική. Οι νέοι κανόνες ε, για τα δημόσια οικονομικά σε ευρωπαϊκό έλεγχο τόνισαν περισσότερο. Ε, εμείς θέλουμε να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τα δύο αυτά, τις δύο αυτές φάσεις, δηλαδή την τεχνική και την κοινοβουλευτική, την ομοθετική και το ελέγχο είναι σημαντικό να επαναλάβουμε την, τον διαχωρισμό ανάμεσα στην αξιολόγηση των δημοσίων δαπανών και την ορθότητα του ελέγχου ε, του εκτελεστικού που ε, επιβαρύνει τους βουλευτές. Έπειτα θα πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητους οργανισμούς από το κυβέρνηση και από το ίδιο το κοινοβούλιο, οπότε σε αυτή την περίπτωση η επεξεργασία των στοιχείων θα πρέπει να ανατίθεται σε εξωτερικούς οργανισμούς. Όμως ο έλεγχος είναι αρμοδιότητα των κοινοβουλίων. ελπίζουμε λοιπόν ότι σύντομα μάλλον θα γίνουν όλα αυτά και στην Ιταλία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Από την Πολωνική Γερουσία, ο κύριος Καζιμίρ Σκλένε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καζιμίρ Σνέινερ, είμαι πρόεδρος ε, της Επιτροπής ε, Ελέγχου του Προϋπολογισμού της ομολογής σας ε, στην Πολωνική Γερουσία. Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη διεξαγωγή και τη διοργάνωση αυτής της συνεδρίασης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Η εκτέλεση του προπολογισμού, οι δαπάνες και ο έλεγχος του προπολογισμού είναι πράγματι αντικείμενο ε, και της βολής και της Γερουσίας μας και προσέχω πάρα πολύ σε αυτά τα θέματα. Στην Βολονία υπάρχει ένας οργανισμός που ασχολείται με τις δαπάνες του προπολογισμού, είναι ένα ανώτατο όργανο, ανεξάρτητη αρχή και έχει ήδη μακρά εμπειρία όσο και παράδοση ε, στον έλεγχο των δημοσίων δαπανών. Παρόλα αυτά, όλο και περισσότερο ε, υπάρχουν αμφιβολίες για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι ότι δεν είναι παρκής. Αυτό το ανώτατο ελεγκτικό όργανο απευθύνεται και στο Κοινοβούλιο και στη Γερουσία ε, και του κάνουμε συστάσεις και το επηρεάζουμε και με μονομένοι βουλευτές, όχι μόνο τα συνολογικά σώματα. Άρα έχουμε και επιρροή στον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος και στους τομείς που γίνεται ο έλεγχος. Βέβαια όλες οι αιτήσει και οι συστάσεις μας δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Είναι και αδύνατο εκ των πραγμάτων έχει έχεις 300-400 βουλευτές ή γερουσιαστές και ο καθένας έχει τις επιθυμίες του. Δεν είναι εύκολο να τα αποκρίνει μέσα στην ίδια χρονιά σε όλα τα αιτήματα αλλά εμείς ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο ελέγχεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού. Η Πολωνική Γερουσία αλλά και η Βουλή ασχολούνται με αυτά τα θέματα και σε ανώτατο επίπεδο, διότι ε, επανειλημμένα κάθε χρόνο η Πολωνική Βουλή λαμβάνει την απαλλαγή. Τώρα τα θέματα του προϋπολογισμού αφορά κυρίως ε, κάποιες άκαμπτες δαπανές, α, συγγνώμη, δαπάνες, δηλαδή που αφορούν κάποιες κοινωνικές δαπάνες, αμοιβές ή εθνικές ε, δαπάνες για την εθνική άμυνα ή ε, ακριβώς δεν έχουμε μεγάλη επιρροή σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση αυτών των δαπανών και δεν υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουμε αυτή, την, αυτή τη διάρθρωση. Πολύ συχνά στη Γερουσία έχουμε ακροάσεις με υπουργούς που μας ενημερώνουν για την ε, πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Πολύ σημαντικό επίσης για μας ε, είναι το γεγονός ότι έχουμε την αίσθηση ότι κάποιες δαπάνες που γίνονται με κοινοτικά κονδύλια δεν είναι πολύ αποτελεσματικές. Γι' αυτό και θα πρέπει να αναλάβουν πολύ σημαντικό ρόλο και οι ελεγκτικοί φορεί τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και οι εθνικοί φορεί ελέγχου για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των κοινοτικών κονδυλίων, ιδιαίτερα του ε, κοινωνικού, Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Δυστυχώ φαίνεται ότι τα κονδύλια του Κοινωνικού Ταμείου δεν είναι πολύ αποτελεσματικά. Υπάρχει πρόβλημα και στην προετοιμασία των προγραμμάτων και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά φυσικά και οι εθνικοί και περιφερειακοί φορείς ε, συμβάλλουν σε αυτήν την αναποτελεσματικότητα. Πολύ ε, ενδιαφέρουσα ήταν η παρουσίαση που μας έγινε από τη Σουηδία για το πώς ε, ετοιμάζει η Σουηδική Βολή τον προϋπολογισμό και πώς εξασφαλίζει την χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Εμείς δεν εφαρμόζουμε ίδιο σύστημα με την Σουηδία, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα το σουηδικό μοντέλο να μας δώσει κάποιες, ε, κάποια τροφή για σκέψη, να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για μας. Γιατί εμείς έχουμε πρόβλημα και στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί και εκεί έχουμε σημαντικά δημοσιονομικά ελλείμματα και στον εθνικό προϋπολογισμό έχουμε εθνικά ελλείμματα. Προσπαθούμε πάντως να τα περιορίσουμε. Βέβαια, η οικονομική κατάσταση της Πολωνίας είναι αρκετά καλή αλλά σίγουρα θα πρέπει να γίνουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις και στην Πολωνία και πολύ ρηξικέλευτες αλλαγές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Μίλτερ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούω τη συζήτηση και εγώ με μεγάλο ενδιαφέρον, ε, όπως και άλλοι συμμετέχω αρκετό καιρό σε αυτή την Επιτροπή και ίσως η πιο κρίσιμη στιγμή ήταν το 1999 όταν για πρώτη φορά μετά από σειρά ετών αρνήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χορηγήσει απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δημιούργησε μεγάλη σύγχυση, συστήθηκε η Ειδική Επιτροπή Σοφών για να εξετάσει με ποιον τρόπο χειρίζεται τα ευρωπαϊκά κονδύλια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκανα την έκθεσή τους αυτή και ένα από τα συμπεράσματα που συγκέντρωσε την προσοχή ήταν ότι είναι δύσκολο να βρει κανείς κάποιον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στα κράτη-μέλη που αισθάνεται πραγματικά την ευθύνη, υπεύθυνο για τη διαχείριση και τις δαπάνες ε, των ε, κοινοτικών κονδυλίων. Ε, στη συνέχεια υποχρεώθηκε σε παρέτηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήρθε η Νέα Επιτροπή πρώτη με νέα συστήματα δημοσιονομικά κτλ. Αλλά έκτοτε Έκτοτε έχουμε δει κάποιες βελτιώσεις, αλλά σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ελεγκτικού συνεδρίου, τα τελευταία χρόνια η κατάσταση επιδεινώνεται. Έχω λοιπόν ε, αυτή τη φράση στο μυαλό μου, ότι είναι δύσκολο να βρεις κάποιον που αισθάνεται υπεύθυνο. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2003 σε κάθε ψήφισμά του για την απαλλαγή αναφέρει ότι χρειάζεται οπωσδήποτε στα κράτη-μέλη που δαπανώνται σε, στην υπευθυνότητα κατά 80% τα κονδύλια να αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη. Γι' αυτό ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπάρχει δήλωση αξιοπιστίας του κράτους μέλους. Δηλαδή κάποιος σε πάση περιπτώσει σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, κεντρικό, ομοσπονδιακό δεν ξέρω αλλά κάποιος πολιτικός ηθήνων να εκδίδει μία δήλωση που να λέγει ότι κατά τη γνώμη του τα χρήματα έχουν δαπανηθεί σωστά ή λάθος εν πάση περιπτώσει, να αναλαμβάνει κάποιο την ευθύνη για αυτά. Στα δικά μα δημοκρατικά συστήματα, Συνήθω όταν κάποιο ψεύδεται ενώπιον ενό κοινοβουλίου ή αλλού, δεν είναι πάρα πολύ καλό για την πολιτική του υγεία στη συνέχεια και ζωή. Και τώρα για δέκατη φορά συναπτή, ε, λέμε ότι κάποιος θα πρέπει να φέρει την προσωπική ευθύνη την πολιτική ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο τα κοινοτικά κονδύλια δαπανώνται στα κράτη-μέλη. Το ξέρω ότι έχουμε ένα νέο δημοσιονομικό κανονισμό που υπάρχει δυνατότητα για πρώτη φορά ένα κράτος μέλος να ε, το κάνει συμμορφούμενο προς τους κανόνες. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να δώσουμε και κίνητρα στα κράτη-μέλη για να το πράττουν. Και έτσι θα έχουν και λιγότερους ελέγχους από τις Βρυξέλλες αν καταλήξουν τα αρμόδια ελεκτικά συνέδρια ότι δαπανώνται καλά τα χρήματα. Θα ήθελα όμως να ακούσω την αντίδρασή σας για αυτή την ιδέα. Ε, πώς γίνεται δεκτή στα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή. Γιατί κατά την άποψή μου δεν πάει άλλο. Δεν μπορούμε για 19η τώρα συνεχή χρονιά να έχουμε ε, ένα ελεκτικό συνέδριο που να μας λέει στην ετήσια έκθεσή του ότι η κατάσταση επιδεινώνεται. Και ενώψη και των ευρωεκλογών δεν είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα, κάτι πρέπει να κάνουμε για να τα βελτιώσουμε. Ευχαριστώ. Ja, vielen Dank, äh, den Kollegen Mulder. Als Ευχαριστώ πολύ. Από την κάτω βουλή των κάτω χωρών θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Έντι Φαν Thank Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε θα ήθελα να απαντήσω και στην έκκληση της κυρίας Γκρέσλε και σε αυτό που ανέφερε τώρα ο κύριος Μιλντερ. Για ποιο λόγο επιθυμώ να το κάνω αυτό, γιατί ανησυχώ πραγματικά για την υποστήριξη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από τους πολίτες για τα κράτη-μέλη, ε, για τα θεσμικά όργανα. Αυξάνεται ο ευρωσκεπτικισμός στις κοινωνίες μας και πιστεύω ότι δεν ισχύει μόνο στην Ολλανδία αυτό και έχει κάποια σχέση μέχρι ενός βαθμού με την αδυναμία μας να απαντούμε με τρόπο ικανοποιητικό για το πώς δαπανώνται τα χρήματα των φορολογουμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι πάρα πολύ επίκαιρη η σημερινή συνεδρίαση και σας συγχαίρω γιατί πραγματικά το θέμα αυτό είναι καυτό. Όπως ήδη ε, τόνισε η κυρία Γκρέσλε, ε, το 80% περίπου του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού δαπανάται σε επίπεδο κράτων μελών, κρατών μελών με συνδιαχείριση. Και μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη-μέλη λοιπόν είναι υπεύθυνα για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι δαπάνες. Το είπε και ο κύριος Μόλντερ αυτό τώρα. Και για 19η συνεχή χρονιά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δίνει αρνητική δήλωση αξιοπιστίας για ε, την διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων. Και αυτό κάπου πρέπει να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν και αυτά τις ευθύνες τους. Συμφωνώ λοιπόν και με την έκκληση του κυρίου Μιλντέρ ότι θα πρέπει κάποιος να είναι υπεύθυνος σε κάθε χώρα και να υπογράφει τις δηλώσεις αυτές γιατί έτσι θα βελτιωθεί και η λογοδοσία Σήμερα λοιπόν θέλω να ρωτήσω και να μάθω αν συμφωνούν με αυτή την ανησυχία συμμερίζονται παρόντες συνάδελφοι και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη λογοδοσία για τη ε, δαπάνη αυτή. Και ένα δεύτερο, μάλλον προτρέχω γιατί αφορά τη δεύτερη ενότητα, είναι το εξή. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε καλύτερη επιτήρηση, εποπτεία ε, στα ποσοστά σφαλμάτων ε, που διαπιστώνονται στα κράτη-μέλη και από τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία τέτοια δυνατότητα. Ευχαριστώ. Να κάνω πρόταση. Έχω άλλους δύο συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο και μετά νομίζω καλό θα ήταν να μπούμε στο δεύτερο τμήμα της συνεδρίασής μας. Από την Ισπανία λοιπόν και την Ισπανική Βουλή θα δώσω το λόγο Στη Γερουσία. Ναι. Ευχαριστώ και καλημέρα σας. Συνεχίζοντας το συνειρμό των προλαλήσαντων, θα ήθελα να πω ότι μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι για 19η συναπτή χρονιά το ελεκτικό συνέδριο δίνει αρνητική δήλωση αξιοπιστίας και επισημαίνει σφάλματα συγκεκριμένων χωρών και δετελεοδεικνύει συγκεκριμένες χώρες όπως η Ισπανία. Εγώ είμαι μέλος της Μεκτής ε, Επιτροπής των δύο σωμάτων της Βουλής ε, που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας ε, των δημόσιων δαπανών. Δεν γνώριζα κάτι τέτοιο. Βλέπουμε ότι ο έλεγχος ε, του δημοσιονομικού ελέγχου του, της Ισπανικής ε, κυβέρνησης, του Ισπανικού κράτους, γίνεται μεταξύ του, ελεκτικού, του Εθνικού Ελεκτικού Συνεδρίου και των τοπικών ελεκτικών συνεδρίων και έχουμε και επίσης τη Μικτή Επιτροπή ε, Βουλής Αντιπροσώπων και Γερουσίας για τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών και των δημοσίων λογαριασμών. Νομίζω ότι ήμασταν πρωτοπόροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί την περασμένη εβδομάδα στην ε, μεικτή αυτή επιτροπή, στην οποία συμμετέχει και ο τη ε, Λόπες, εγκρίναμε την ίδρυση μιας ανεξάρτητης αρχής ε, δημοσιονομικής ευθύνης για να ελεγχθεί η συμμόρφωση σε ό,τι αφορά τα όρια του με τον περιορισμό, τα όρια του περιορισμού των δαπανών και του περιορισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος και της σωστής αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων. Και με την παρουσία του Υπουργού Μοντόρο που είχε προσκληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δώσει λόγια το υψηλό ποσοστό σφάλματος, πιστεύω ότι με όλα αυτά τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες θα πολλές, θα διασκεδαστούν πολλές αμφιβολίες ό,τι αφορά την, τις παρατυπίες που διαπιστώθηκαν στην ισπανική διαχείριση των κοινοτικών κονδύλων, κυρίως του Ταμείου Ανάπτυξης. Ευχαριστώ και τελευταίος ο ε, σε αυτό τον πρώτο γύρο, το Εθνικά Κοινοβούλια, ο συνάδελφος του το Καμπρίτα από την Πορτογαλική Βουλή. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω τη σημασία αυτής της ε, ε, συνάντησης εδώ, γιατί υπάρχουν μεγάλες αμφιβολίες για το ευρωπαϊκό σχέδιο, γιατί τα προβλήματα τα οικονομικά βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού και της συζήτηση σε διεθνές επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή συζήτηση όσον αφορά την καλή διαχείριση και έλεγχο της χρήσης των δημοσίων δαπανών ε, και επίσης την, τον ελεγκτικό ρόλο των εθνικών Ευρωπαϊκού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία όσον αφορά την προσοχή και τη σημασία που έχει η δημόσια συζήτηση όσον αφορά τι αλλαγέ και τι μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν ε, στο μέλλον. Γίνεται, δίνεται δε και λίγο μικρότερη προσοχή στους, προπολογισμού, ε, μάλλον μεγαλύτερη προσοχή από την παλιότερα, στο πώς ακριβώς ε, καταρτίζονται και πώ εκτελούνται οι προπολογισμοί καθώ και αν ανταποκρίνονται στου στόχου που αρχικά είχαν τεθεί. Θα πω ότι στην Πορτογαλία λόγω γενικών συνθήκων αλλά και λόγω συγκυρίας, γιατί είναι μια χώρα που περνά μια πολύ δύσκολη διαδικασία δημοσιονομικής εξυγίανσης, το θέμα είναι ότι το θέμα, ότι το ζήτημα του προπολογισμού, των δημοσιονομικής εξυγίανσης είναι στο επίκεντρο της συζήτησης σε όλη τη χώρα αλλά και στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω για το ποια είναι η μορφή που με την οποία, ποιος είναι ο τρόπος μάλλον με τον οποίο εμείς ε, παρακολουθούμε και συζητούμε τα θέματα τα δημοσιονομικά. Ο προϋπολογισμός ε, ε, δημοσιεύεται σε μια έκθεση που συντάσσεται από το Κοινοβούλιο και, εκδίδεται από το Κοινοβούλιο τριμενιαίως κάθε τρει μήνες δηλαδή, ε, και γίνεται συζήτηση στο Κοινοβούλιο ανάμεσα στην Επιτροπή Οικονομίας και την Κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο ε, θα εκτελεστεί ή εκτελέστηκε μάλλον ο προϋπολογισμός. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον ανεξάρτητο τώρα έλεγχο γίνεται από το Κοινοβούλιο ε, σύμφωνα με το σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου και τον ΙΠΑ όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, ε, το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο δημιούργησε μία ειδική επιτροπή τεχνικής υποστήριξης με ανεξάρτητους συμμετέχοντες που λειτουργεί ταυτόχρονα με την Επιτροπή Δημοσιονομικού και, Προπολογισμού και Οικονομίας και συζητά τα θέματα τα δημοσιονομικά αλλά και τα θέματα δημοσίου ελλείμματος. Τρίτο επίπεδο ελέγχου το Κοινοβούλιο πέρασε ε, τις αρμοδιότητες του και ζήτησε τέσσερις ελέγχους συγκεκριμένους. Δύο που γίνονται από το ελεκτικό συνέδριο όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες. Δύο γίνονται από το ελεκτικό συνέδριο και άλλες δύο από τα, ε, ε, τα ιστορικά έργα ελέγχου θα εξαρτώνται από την κυβέρνηση. Εν τέλει, όσον αφορά την εθνική διάσταση, όσον αφορά δηλαδή τους γενικούς λογαριασμούς του κράτους και το Δικαστήριο ε, Δημοσίων Δαπανών, Δημοσίων μάλλον Λογαριασμών, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ε, αυτό υποβάλλει τις ε, απόψεις του για το γενικό κατάσταση των λογαριασμών του κράτους, υποβάλλει συστάσεις για θέματα επιτυχίες που πρέπει να αλλάξουν τόσο όσον αφορά τους, δημο, τους δημοσιονομικούς ελέγχους αλλά και όσον αφορά την κατάρτιση του προϋπολογισμού και ε, προβαίνουμε έτσι σε νομοθετικά, νομοθετικές προτάσεις σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Και τέλος ε, και χαιρετίζω και το δόκτωρα Βιτάλ Καλντέιρα που είναι ο εκπρόσωπος της Πορτογαλίας στο Ελεκτικό, Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο και γίνεται λοιπόν τακτικά μια έκδοση ε, που αναφέρει τη, ε, τις εξελίξεις κάθε φορά για τον προϋπολογισμό και είναι το βασικό, η βασική συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομίας και Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου αλλά και στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έτσι ώστε να γίνεται ε, ο έλεγχος όσον αφορά τη διαχείριση των εθνικών αλλά και των ευρωπαϊκών πόρων. Πάντως ένας ορθός έλεγχος των δημοσίων δαπανών υποχρεώνει στο να είμαστε αποτελεσματικοί θα πρέπει να βρούμε δομής προτεραιότητας και να ορίσουμε είτε είναι μεγάλες επενδύσεις, είτε είναι η στήριξη στις πολιτικές απασχόλησης, τη γεωργία, οι δραστηριότητες μπορεί να ποικίλουν από χώρα σε χώρα, πάντως να υπάρχει μια επιλογή, γιατί προσπαθώντας να κάνουμε πως θα ελέγχουμε όλα, ε, ο κίνδυνος είναι τελικά να μην ελέγχουμε αποτελεσματικά τίποτα. Κάτι ακόμα σε σχέση με τα στοιχεία που έδωσε ο συνάδελφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το τις χώρες όπου υπάρχουν πιο πολλές ε, ε αντικανονικότητες. Ε, εγώ πιστεύω πως θα πρέπει να, να, βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της ανάλυσής μας και την ορθότητα αυτής, καθώς και την αποτελεσματικότητα των δαπανών. Δεν αρκεί να επαληθεύουμε αν, έγινε, αν υπήρξαν ή όχι αντικανονικότητες ή προβλήματα. Θα πρέπει ε, να δούμε αν οι δαπάνες που έχουν αφιερωθεί για τα ευρωπαϊκά προβλήματα προγράμματα ή για τις πολιτικές απασχόλησης, αν ε, αυτές ε, τελικά επέτυχαν τους στόχους και τις προσδοκίες τους εθνικούς, τους ευρωπαϊκούς, αλλά και κυρίως τις προσδοκίες των, κρατών, των, των πληθυσμών μας, των λαών μας, που αυτοί μας δίνουν ε, την έγκριση για να μπορούμε και εμείς να κρίνουμε αυτές τις δαπάνες. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Πολύ ζωντανή η τοποθέτηση και πολύ σχηδής. Μας παρουσιάσετε πολλά θέματα όλοι ε, στην πρώτη ενότητα του πρωινού μας. Κλείνει λοιπόν εδώ, αν μου επιτρέπετε, και ε, θα ακούσουμε τώρα την παρουσίαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λεκτικού Συνεδρίου, του κύριο Καλτέρα. Σας καλωσορίζω θερμότατα σε αυτή τη διακοινοβουλευτική διάσκεψη. Θα ήθελα και πάλι να τονίσω αυτό που είπε ο συνάδελφος Καπρίτα και άλλοι είναι σημαντική τούτη εδώ η συνεδρίαση από τη σκοπιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι επιτροπές ε, ελέγχων των προπολογισμών αλλά και οι επιτροπές προπολογισμών των κοινοβουλίων των κρατών μελών να ανταλλάζουν απόψεις και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αναπτύξουμε μια συναντήληψη για το τι σημαίνει χρηστή ε, εκτέλεση του προπολογισμού και καλή διαχείριση. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε τόσους πολλούς συναδέλφου από τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, τεχνικώ θέλω να σα πω το εξή. Στη δεύτερη ε, ενότητα ε, οι σελίδε που σα έχουν διανεμηθεί για να δείξω το λόγο έχουν χρώμα πορτοκαλί. Στο πρώτο ήταν πράσινο, τώρα τελείωσε αυτό και τώρα πάμε στο πορτοκαλί. Διευκολύνει και τη γραμματεία αυτό για να έχει μια εποπτεία και στα τυπικά θέματα και τα διαδικαστικά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας δώσω το λόγο κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Τόιερ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Κυρίες και κύριοι, με τιμά ιδιαίτερο η πρόσκλησή σα ε, στη συνεδρίαση αυτής της Διακοινοβουλευτική Επιτροπής με θέμα τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών που είναι σημαντικό στοιχείο της υποχρεώση λογοδοσία. Ο έλεγχος του κοινοτικού προϋπολογισμού αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση πολλό δε μάλλον που το 80% των ε, κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εμπίπτουν στην επιμερισμένη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω κάποιες παρατηρήσεις ε, σε σχέση με την πρόκληση αυτή υπό το πρίσμα του Ελεκτικού Συνεδρίου που είναι το θεσμικό όργανο το αρμόδιο για τον έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να καλύψω ορισμένα θέματα όπως ε, πώς θα καταφέρουμε αποτελέσματα επιτόπου, πώς θα μειώσουμε το γραφειοκρατικό άχθος και το διοικητικό άχθος, πώς θα καταστήσουμε πιο αποτελεσματικό τον έλεγχο και το δημοσιονομικό έλεγχο, θα βελτιώσουμε τη την διαφάνεια, ιδιαίτερα για τις δαπάνες της συνοχής και της γεωργίας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πού δαπανώνται τα χρήματά τους, κατά πόσο αυτά δαπανώνται σωστά και αν πραγματικά πιάνουν τόπο σε ό,τι αφορά το λογαριασμό της Ευρωπαϊκής, τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, να διαβεβαιώνονται για την αξιοπιστία των δημοσίων λογαριασμών, των ενωσιακών λογαριασμών, για την ε, χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Αυτό άλλωστε απαιτούν και οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για η χορήγηση τέτοιων ε, εχεγγύων όμω ε, στου Ευρωπαίου πολίτε δημιουργούνται τεράστιε προκλήσει για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη. Σημαντική πρόοδο έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά δυστυχώ έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε μέχρι ότου διαβεβαιώσουμε πλήρους του Ευρωπαίου πολίτε για όλα αυτά τα θέματα. Αυτό είναι το μήνυμα και τη ετήσια έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2012 που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Η έκθεση κάνει μια γενική επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης ε, της ε, δημοσιονομικής διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν ολίγης, η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ελεκτικού Συνεδρίου για το 2012 ε, λέει «Γνωρίζουμε σε τι δαπανώνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπονούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αξιόπιστοι ε, κάτι που ισχύει από το 2007. Γνωρίζουμε βέβαια ότι δεν αξιοποιούνται σωστά όλα τα κονδύλια. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δυστυχώς υπάρχει ποσοστό σφάλματος στους ε, λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα το ποσοστό αυτό σφάλματος ανέρχεται στο 4,8% για το 2012, αλλά δεν γνωρίζουμε αρκετά στοιχεία για την συνολική αξία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί τα, τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν δίνουν επαρκείς ε, ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες για τα αποτελέσματα της ε, δαπάνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ε, κάποιε ελλειπεί γνώσει ό,τι αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο του ευρωπαϊκού προπολογισμού και γίνονται τεράστιε προσπάθειε για τη βελτίωση αυτών των αδυναμιών τα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνεργάζεται με ένα ευρύτερο φάσμα εθνικών αρχών προκειμένου να γίνει καλύτερη διαχείριση και έλεγχο των κοινοτικών κονδύλιων. Μία επιπλέον πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να εξασφαλίσει ότι αυτές οι ρυθμίσεις για τη διαχείριση και τον έλεγχο των κοινοτικών δαπανών ευθυγραμμίζονται με τις ε, ρυθμίσεις για τον εξωτερικό δημοσιονομικό έλεγχο και, το, και την πολιτική εποπτεία που προβλέπονται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για να εξασφαλίσει η διαβεβαίωση στους Ευρωπαίους πολίτες ε, για τη χρηστή διαχείριση θα πρέπει να έχουμε συνάρθρωση τριών επιπέδων και στρωμάτων του, του επίπεδου της ε, διαχείριση και ελέγχου, του επίπεδου του εξωτερικού δημοσιονομικού ελέγχου και του επίπεδου της πολιτικής εποπτείας. Όλοι αυτά τα επίπεδα θα πρέπει να συνδυάζονται. Αν θέλουμε αποτελεσματικό και αποδοτικό δημοσιονομικό έλεγχο και μία πολιτική εποπτεία, θα πρέπει να ξεκινήσουμε με την θέσπιση αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου. Έχουμε βελτιώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ε, διάφορες αυτές ρυθμίσεις και από το 2004 εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο εσωτερικό σύστημα και πλαίσιο ελέγχου για τον έλεγχο των κοινοτικών κονδυλίων στα κράτη-μέλη. Και μάλιστα το ελεκτικό συνέδριο είχε υποβάλει μια σχετική πρόταση το 2002 στην γραμματότηση για το ενιαίο ε, ελεκτικό μοντέλο. Ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός προβλέπει κάποια ε, κάποιες απαιτήσει ότι αφορά τις, ε, τις που θα πρέπει να δίνουν τα κράτη-μέλη στις ε, εθνικές δηλώσεις τους αξιοπιστίας. Και επίσης θα πρέπει αυτές οι διαβεβαιώσεις να χρησιμοποιούνται για τις εθνικές, συστάσεις, τις εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας για τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να βελτιώσει την νομοτυπία και την κανονικότητα των πληρωμών γίνεται προσπάθεια να μειωθεί το επίπεδο των παρατυπιών κάτω από το 2% προκειμένου να εξασφαλιστεί θετική δήλωση αξιοπιστίας από το ελεκτικό συνέδριο. Δυστυχώς αυτός ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί ακόμη. Το ελεκτικό συνέδριο προβλέπει ότι από το 2007 είχαμε σημαντική μείωση του ποσοστού σφάλματος. Δυστυχώς όμως υπάρχει ακόμη ένα αισθητό ποσοστό σφάλματος και μάλιστα τα τελευταία τρία χρόνια είχαμε και μια αύξησή του. Τα περισσότερα σφάλματα εντοπίζονται στο 80% του κοινοτικού προπολογισμού που ε, αφορούν κονδύλια της συνοχής και της γεωργίας ε, για τα οποία ισχύει επιμερισμένη διαχείριση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών. Θα πρέπει και οι εθνικές και περιφερειακές αρχές ε, να, να προλαμβάνουν και να εντοπίζουν καλύτερα τα σφάλματα. Γι' αυτό θα πρέπει να βελτιωθούν οι εσωτερικοί έλεγχοι που μέχρι στιγμής είναι μερικώς μόνο αποτελεσματικοί. Επίσης, οι δοκιμές εναλλαγών που κάναμε στο ελεκτικό συνέδριο κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα ποσοστά σφάλματος θα έπρεπε να ελέγχονται και να διορθώνονται από τις εθνικές αρχές πριν υποβληθούν οι αιτήσει για επιστροφές δαπανών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα τμήμα του προβλήματος ε, οφείλεται στο γεγονός ότι το ισχύον σύστημα ε, δημοσιονομικών διορθώσεων ε, δεν επιτρέπει, δεν ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να διορθώσουν ή να αποτρέψουν τα λάθη προκειμένου να φτάνουν τα κονδύλια στους πραγματικούς και επιλέξιμους δικαιούχους. Αλλά και οι κανόνες δαπανών ε, φέρουν την ευθύνη σε κάποιο βαθμό για τα λάθη. Μερικές φορές είναι υπερβολικά περίπλοκοι αυτοί οι κανόνες. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις δαπάνες ε, ε, επικεντρώνεται κυρίως στην κατανομή των δαπανών και, στην, και στην, στον επιμερισμό των κονδυλίων και όχι στην ενθάρρυνση της επιδίωξης αποτελεσμάτων. Υιοθετούμε λοιπόν στο ελεκτικό συνέδριο μια διαφορετική προσέγγιση. Μια προσέγγιση που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην προώθηση της απόδοσης των καλύτερων επιδόσεων. Θέλουμε πιο αποτελεσματική δαπάνη. Κατά τη γνώμη μας, ποιοτικέ δαπάνες ε, θα πρέπει να σέβονται τους κανόνες και ταυτόχρονα να υλοποιούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Τα προγράμματα δαπανών θα πρέπει να εκπληρώνουν όλους αυτούς τους στόχους τη διαφάνεια, τη λογοδοσία ε, και επίσης οι ρυθμίσεις ελέγχου θα πρέπει να καλύπτουν και τις δύο αυτές πτυχές. Κάτι που προβλέπει αναθεώρηση των κανόνων διαχείρισης και ελέγχου προκειμένου να δοθεί περισσότερη έμφαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Μέχρι στιγμής ε, οι κανόνες αυτοί κυρίως ε, επικεντρωνόταν στην ομοτυπία και την κανονικότητα των πληρωμών το, ο, η περίοδος προγραμματισμού 2014-2020 μας δίνει μία μοναδική ευκαιρία για την βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των κοινοτικών δαπανών. Μετά από εκτενείς συζητήσεις θα εθετηθούν ε, οι βασικές νομοθετικές προτάσεις για τα προγράμματα δαπανών και το νέο, υπό το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Την επόμενη επταετία γύρω στα 800 δισεκατομμύρια ευρώ θα δαπανηθούν με βάση την επιμερισμένη διαχείριση για τη συνοχή και τη γεωργία. Το ελεκτικό συνέδριο έχει ε, δώσει πολλές ε, γνωμοδοτήσεις για τη βασική νομοθετική διαδικασία. Φαντάζομαι τις γνωρίζετε. Κατά την άποψη του ελεκτικού συνεδρίου, μερικές ε, ευκαιρίες για την απλοποίηση των κανόνων και τη βελτίωση των προγραμμάτων δαπανών δυστυχώς έχουν ήδη χαθεί. Σε ό,τι αφορά τη συνοχή, πολλά θεμελιώδη στοιχεία αυτών των προγραμμάτων ε, ρυθμίζονται σε μεταγενέστερο στάδιο και σε υποδέστερο επίπεδο με εφαρμοστικές και κατεξουσιοδότηση πράξεις. Βέβαια είναι σαφές ότι το συνολικό νομικό πλαίσιο εξακολουθεί να παραμένει περίπλοκο. Προβλέπονται έξι επίπεδα κανόνων και σε μερικές περιπτώσεις ένα πρόσθετο έβδομο επίπεδο της εθνικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, το Ελεκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι το διοικητικό άχθος για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τις εθνικές θα παραμείνει υψηλό. Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για τη διαχείριση και τον έλεγχο, το ελεκτικό συνέδριο χαιρετίζει το δυναμικό απλούστευση των κρατών μελών για τα διαχειριστικά προγράμματα. Θεωρεί όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, διαδραματίσει πιο ενισχυμένο ρόλο στην πιστοποίηση των εθνικών διαχειριστικών αρχών και στον έλεγχο της αξιοπιστίας του έργου των ελεκτικών αρχών. Κατά τη γνώμη μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μέτρα για την εξασφάλιση του, της ποιότητας του ελέγχου των δηλώσεων αξιοπιστίας των εθνικών αρχών και τις πληροφορίες για την εκτέλεση των, προβλημάτων, προγραμμάτων. Αυτή η ενημέρωση και η δήλωση αξιοπιστίας θα πρέπει να είναι σημαντικής ποιότητας και να πληρεί τις ανάγκες ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Δυστυχώς ε, εξακολουθούμε να επικεντρωνόμαστε στις εισρωές. Ε, έχω, έχει χαθεί σημαντική ευκαιρία να στοχεύσουμε και να προσανατολίσουμε τα προγράμματα προς τα αποτελέσματα. Θα πρέπει να έχουμε σαφέστερους στόχους, κατάλληλους δείκτες, στενότερη σύνδεση πληρωμών και αποτελεσμάτων και καλύτερες και πιο αυστηρές απαιτήσει για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της απόδοσης σημαντικά στοιχεία θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω για να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας προσανατολισμένης προς την απόδοση. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει την εισαγωγή εθνικών συμβάσεων εταιρική σχέση, νέων πλαισίων απόδοση και αποθεματικών απόδοση. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε την ε, εισαγωγή αυτών των νέων στοιχείων στι ε, ισχύουσε ρυθμίσει διαχείριση και ελέγχου. Σε ό,τι αφορά την κοινή γεωργική πολιτική, το ελεγκτικό συνέδριο έχει παρόμοιες απόψεις για την περιπλοκότητα του νομικού πλαισίου, την αυξανόμενη χρήση κατεξουσιοδότηση και εφαρμοστικών πράξεων, την ανάγκη της ενίσχυσης του υποπτικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την υπερβολική έμφαση που δίνεται στις ροές αντί για τα αποτελέσματα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατρέχει κίνδυνο. Αν οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, πρέπει να πιστούν για την ανάγκη των ε, ευρωπαϊκών, των ενωσιακών προγραμμάτων πρέπει να είναι βέβαιοι για, την προστιθέμενη αξία αυτών των προγραμμάτων. Θα πρέπει να καθησυχάσουμε τους πολίτες ε, και να τους διαβεβαιώσουμε ότι τα κοινοτικά κονδύλια αξιοποιούνται με σωστό τρόπο και χάνουν χρηστή διαχείριση. Αλλά κάτι τέτοιο δεν αρκεί. Να σα δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Δεν αρκεί οι πολίτε να γνωρίζουν ότι θα κατασκευαστεί ή θα εξυγχρονιστεί ένα θαλάσσιο λιμένα, ότι χτίζονται αποθήκε και αποβάθρε. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτε ότι αυτέ οι ε, δυνατότητε αξιοποιούνται. Θα ελιμενίζονται και αγκυροβολούν λιμάνια, ε, πλοία συγγνώμη, στα λιμάνια. Έχουμε μεταφορά των φορτίων από τα λιμάνια στο σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο και δημιουργούνται θέσει απασχόληση. Τέτοια αποτελέσματα περιμένουν οι πολίτε κάτι τέτοιο μας φέρει να ελέγξουμε τα όρια του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και μάλιστα με κοινό τρόπο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και με κατάλληλη υποπτία. Όταν τα εθνικά και τα ενωσιακά κονδύλια δαπανούνται από κοινού θα πρέπει ο εθνικός έλεγχος ε, να εξασφαλίζεται σε επίπεδο εθνικό, αλλά να ε, γίνεται και ευρωπαϊκός έλεγχος από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να διαθετήσουμε μια διτή προσέγγιση για να προωθήσουμε τη χρηστή διαχείριση και την καλύτερη δαπάνη. Θα πρέπει, δεδομένες και της κρίσης, να έχουμε πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα με λιγότερα κονδύλια, άσχετα αν τα κονδύλια είναι εθνικά ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης, αλλά και της λογοδοσίας. Και φυσικά με τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε μέτρα ώστε να γίνει με εναρμόνιση των ε, δημοσιονομικών και ελεκτικών πλαισίων των δημοσίων φορέων των κρατών μελών. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα θεσμικά όργανα ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο αλλά και τα Εθνικά Ελεκτικά Συνέδρια θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο προκειμένου να δημιουργηθούν θετικές εξελίξεις στη δημοσιονομική διαχείριση και στον έλεγχο τα επόμενα χρόνια ώστε να εξασφαλίσουμε καλύτερη ε, και ε, μεγαλύτερη αξιοποίηση των δημοσίων δαπανών χάρη των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ, ήταν ιδιαίτερη τιμή η συμμετοχή μου σε αυτή τη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Καλτέρα για την εισαγωγή σας στη δεύτερη ενότητα της σημερινής συνεδρίασης. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Μεν Χάιντερ, ε, μέλος της Αυστριακής Βουλής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ είμαι. Κυρίες και κύριοι, ε, αναφέρθηκε πολλές φορές το θέμα της αναγνώρισης Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αποτελεσματικής ή αποτελεσματικότερης χρήσης των δημοσίων κονδυλίων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αλλά προϋποθέτει και αποτελεσματικό έλεγχο. Οι εξελίξεις τα τελευταία χρόνια κατέδειξαν ότι είναι επιγόντως απαραίτητο να ξαναδούμε την αρχιτεκτονική του ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τη βελτιώσουμε. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι και ακριβώς η ε, έλεγχη ε, για το σκόπιμο κάθε έργο, για ε, το νομότυπο και το αναλογικό. Δεν αρκεί να το κάνει αυτό μόνο το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο και επίσης δεν αρκεί για να ε, εφαρμόζονται σωστά οι νέες οδηγίες και οι νέοι κανονισμοί. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνονται παντού έλεγχοι ε, και ε, γι' αυτό μιλώ για την αρχιτεκτονική των ελέγχων και συστηματική έλεγχη τα εθνικά κοινοβούλια και κυρίως τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια ε, που είναι ελεγκτικοί οργανισμοί έχουν και γνώση και εμπειρία στην οποία μπορούμε και πρέπει να ανατρέχουμε. Η απαραίτητη μεταξέλιξη λοιπόν της αρχιτεκτονικής των ελέγχων θα πρέπει να βασίζεται και στην εμπειρία και τη γνώση των εθνικών ε, ελεκτικών συνεδρίων. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται λοιπόν στη διαδικασία της εκπόνησης των νέων μηχανισμών ελέγχων ακριβώς λόγω της παράδοσης της εμπειρίας και της γνώσης τους. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, τον συνάδελφο Χάιντερ από την Αυστρία. Δεν έχω άλλους συναδέλφους να έχουν ζητήσει το λόγο από τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρία Γκρέσλε. Ναι. Όπως πάντα, εδώ πέρα ορκιζόμαστε ο ένας τον άλλον αιώνια φιλία. Αλλά επί της ουσίας τι κάνουμε και θέλω να ρωτήσω τη Λουθουανή συνάδελφο. Μέχρι τώρα τι έχετε κάνει για να αντιμετωπίσουμε το προβληματικό παιδί ε, <laughs> στη Λιθουανία που είναι το πυρηνικό εργοστάσιο της Ιγναλίνα. Ξέρουμε πως έχει κατάσταση, είχαμε μεταβεί εκεί, δεν θυμάμαι αν ήταν το 11 ή το 12 και ε, σας ερωτώ Πώς παρακολουθείτε αυτή την υπόθεση της ε, Ιγναλίνα. Ε, έχουμε συγκρουστεί επανειλημμένα με την κυβέρνηση της Λιθουανίας. Κάπως έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Να ρωτήσω και τον Ιταλό συνάδελφο τι προτίθεστε να κάνετε για να σταματήσει αυτή η ηγετική θέση που έχει η Ιταλία στα σφάλματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στο Λάκυλα τι έγινε. Θυμάστε εκεί που έχει γίνει ο σεισμός και λυπούμεθα πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά όταν είναι μια σεισμογενής περιοχή και μετά από ένα σεισμό είναι τεράστια τα προβλήματα. Εσείς πώς παρακολουθείτε τις δαπάνες του Ιταλικό κράτος. Τα κοιτάτε αυτά, τα εξτάζετε. Παρακαλώ συγκεκριμένες απαντήσεις για να συζητάμε σε γερό έδαφος και όχι απλές προθέσεις ε, και εξαγγελίες να δηλώνουμε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Γκρέσλε. Τώρα δεν ξέρω αν θέλουν να απαντήσουν οι συνάδελφοι. Είναι ε, στη διακριτική του ευχαίρεια. Υπεχρεωμένοι δεν είναι όπω θέλουν. Παρακαλώ, η κυρία Βαϊκιέν. Σα ευχαριστώ για την ερώτησή σα, κυρία Γκρέσλε. Έχουμε δημιουργήσει μια κοινοβουλευτική επιτροπή των ε, ενεργειακών ε, υποθέσεων και ασχολείται με, αυτή, με αυτό το πυρηνικό σταθμό. Επίσης ασχολείται με το θέμα το Υπουργείο Οικονομικών. Ε, ε, αυτή τη στιγμή έχουμε ολοκληρώσει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών για να δούμε δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να, θέσουμε σε, να υλοποιήσουμε το σχέδιο. Θα έλεγα ότι θα ήθελα μάλλον να προσθέσω ότι σε όλα τα επίπεδα στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο είναι ένα θέμα ε, πάρα πολύ σημαντικό και προσπαθούμε να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Θέλουμε να το φέρουμε σε αίσιο πέρα. Σε ευχαριστώ. vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια θα ήθελα να δώσω το λόγο στο συνάδελφο από την Ιταλία. Ο κύριος Καριέλο. Ευχαριστώ. θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον Πρόεδρο Καλντέρε για την ε, εισήγησή του που τόνισε τις, ε, τη σημασία των λειτουργιών του εξωτερικού ελέγχου όσον αφορά τις ε, δαπάνες. Και εκμεταλλεύουμε την ευκαιρία για να απαντήσω σε σχέση με τα όσα ανέφερε η κυρία Γκρέσλεφ. Το Κοινοβούλιο σίγουρα θα μπορούσε να αναλάβει μια ερευνητική ε, και αναγνωριστική ε, υπόθεση ε, γιατί αυτά έγιναν στην περασμένη θητεία αλλά σε αυτήν την, εδώ την σημερινή συνεδρίαση θα ήθελα να υπογραμμίσω τις δηλώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της ανάλυσης εκείνης της έκθεσης από τον ίδιο τον Επίτροπο Χάν και τον Γενικό Διευθυντή της DG Regio της, Γενικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Πόπενσε. Σε εκείνη την αξιολόγηση λοιπόν είχε ήδη υπογραμμιστεί πως ε, το υπερβολικό κόστος ε, των ε, καταλήμματων σε σχέση με μια κανονική φυσιολογική υγεία καθορίστηκε κυρίως από τον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης και από το γεγονός ότι χρειαζόταν να εξασφαλιστεί στέγαση επιγόντως για πάνω από 10.000 ανθρώπους που είχαν εκτοπιστεί θύματα του σεισμού στο Αμπρούτσο. Άρα λοιπόν η ρυθμή εργασίας 24 ώρες 24ωρο αλλά και τα κριτήρια κατασκευής, τα αντισυσμικά, που καθορίζονται από την ε, περιοχή αναφοράς ε, οδήγησαν σε αύξηση του κόστους. Αυτές είναι εκτιμήσεις που προέρχονται από την ε, τρέχουσα θητεία που μπορεί όμως να αναλάβει και εμβάθυνση της έρευνας στο θέμα. Πάντως ήδη υπάρχει αξιολόγηση και μάλιστα τεκμηριωμένη που έχει θεμελιώσει αυτές τις θέσεις. Κατά τη γνώμη μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά να αναλάβω την δέσμευση να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες ίσως στο μέλλον. Θεωρώ πάντως πως είναι σε αυτή τη φάση σημαντικό να σας ενημερώσω για την ε, Ιταλική προσέγγιση σε σχέση με τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων όπως την έχει διαμορφώσει ο Υπουργός ε, Ορμόδιο. Εμεί θεωρούμε πω είναι καλύτερη πρόληψη από τη θεραπεία και γι' αυτό το, Ευρωπαϊκό, το Ιταλικό Κοινοβούλιο εν ώψη τη επόμενη προγραμματικής περίοδου 2014-2020 προβλέπει ενίσχυση των μέσων που επιτρέπουν να προληφθούν οι παρατυπίε και οι ανεπάρκειε στη δαπάνη των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων. Η πιο σημαντική περίπτωση είναι η πρόσφατη απόφαση που ελήφθη όντω από τον Υπουργό για τη δημιουργία ενό οργανισμού με αρμοδιότητες στήριξης στη φάση προγραμματισμού και της διαχείρισης από την πλευρά ε, των ε, των ε, ελέγχων, γιατί η διαχείριση θα πρέπει να ελέγχεται όχι μόνο από κεντρικό επίπεδο, αλλά και στις ίδιες τις περιφέρειες. Με τη δημιουργία αυτού του οργανισμού που θα συζητηθεί μέσα στο πλαίσιο του νόμου περισταθερότητας, για να μπορέσουμε να προλάβουμε τα σφάλματα που έγιναν την περίοδο 2007 και 2003 που, που τη δυνατότητα να δαπανηθούν οι πόροι που, είχαν, που αναλογούσαν στην Ιταλία στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων. Να θυμίσω ότι δύο χρόνια πριν από την τελική προθεσμία για την ε, εκπνοή της προθεσμίας ε, για την επαλήθευση των ε, δαπανών, δυστυχώς οι δαπάνες ανέρχονται μόλις σε 19 ε, λίγο παραπάνω δηλαδή από το 40% των προγραμματισμένων δαπανών. Η δημιουργία αυτού του οργανισμού λοιπόν στόχο έχει να ζητήσει, ε, να προσπαθήσει να, να δαπανίσει τα χρήματα με τον καλύτερο, το πιο διαφανή και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και ταυτόχρονα να προλάβει ενδεχόμενα σφάλματα στην διαχείριση αλλά και στην μεταφορά στοιχείων αλλά και στη χρήση των κονδυλίων. Άρα λοιπόν η στήριξη της οργανισμού προς τις περιφέρειες θα πρέπει να βελτιώσει τη δυνατότητα προγραμματισμού και δαπάνες με κατάλληλο τρόπο για όλα τα κονδύλια που προβλέπονται από το πρόγραμμα 2014 με 2020 προβλέποντας, όπως είπα, και προλαμβάνοντας κάθε παρατυπία. Επίσης ε, θέλουμε να επιβάλλουμε μια εξάντε παλήθευση, δηλαδή κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορούν να είναι καν υποψήφιες οι περιφέρειες για, ε, για να πάρουν ε, κονδύλια. Και επίσης να υπάρχουν και ρυθμίσεις κυρώσεις όσον αφορά την ελλειπή εφαρμογή η δαπάνη, ελληματική δαπάνη των κονδυλίων. Θα ήθελα επίσης να ε, πω τα εξής όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν από το να συνέδριο όσον αφορά την ε, ε, τυπικότητα αλλά και την ε, αποτελεσματικότητα της δαπάνης και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Γίνεται σημαντική συμβολή στον έλεγχο ε, με αυτόν τον τρόπο ε, από πλευρά του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου γιατί δημιουργείται και ένα κοινοβουλευτικό γραφείο για τα δημοσιονομικά θέματα που θα ελέγχει τα στοιχεία και μακροοικονομικά. Ωστόσο δεν μπορώ να κρύψω σε σχέση με την Ιταλική εμπειρία πως το Κοινοβούλιο δεν έχει πάντοτε τα μέσα και τις δυνατότητες αλλά και την ε, πολιτική βούληση κάποιες φορές να παρέμβει ή να δώσει συνέχεια στα όσα ε, ε, αναφέρει το Ελληνικό Συνέδριο. Αναφέρομαι δηλαδή στην μεγαλύτερη υπευθυνότητα που απαιτείται από, αυτήν την, από αυτό το σώμα. Κάποιες φορές μάλιστα φτάνουμε σε κάποια απόσταση από σε παράνομες και παράτυπες ε, ε, λειτουργίες. Ε, ίσως ορισμένα κανάλια μπορεί να έχουν καθορίσει και στην απόρριψη των ευθυνών, γιατί αυτό μπορεί να συνδέεται και με παρανομίες. Ε, θα πρέπει δηλαδή να βελτιώσουν οι χρόνοι, οι προθεσμίες ε, ανάμεσα στις οποίες φτάνουν κάποιες εκθέσεις ε, και μετά τις αναλαμβάνει και τις εκπαιδεώνει το Κοινοβούλιο ώστε το Κοινοβούλιο να αναλάβει και εκείνος, εκείνο εγκαίρος της ευθύνης του, την κατάλληλη στιγμή δηλαδή. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Ιταλό συνάδελφο για τις ε, διευκρινήσεις που έδωσε και τις απαντήσεις στην κυρία Γκρέσλε. Θα ήθελα να πω ότι η συζήτηση αυτή δεν περιορίζεται στην Ιταλία. Πολλές χώρες, ακόμη και η Δανία, είχαν προβλήματα στην ε, εκτέλεση των κοινοτικών κονδυλίων. Δεν είναι ιδιαίτερο πρόβλημα της Ιταλίας. Απλώς η Ιταλία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δούμε πώς χρησιμοποιούν οι εκθέσεις του ελεκτικού συνεδρίου στα εθνικά κοινοβούλια. Γιατί στα τέλη του 2012 το ελεκτικό συνέδριο εκπώνησε ειδική ε, ενδελεχή έκθεση για το σεισμό στην Άκουιλα και ε, θα ήθελα να ρωτήσω τον Ιταλό συνάδελφο αν η σχετική έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου εξετάστηκε στην ε, Ιταλική Βουλή ή σε κάποια από τις ειδικέ επιτροπές ε, της Ιταλικής Βουλής. Γιατί από τη στιγμή που δόθηκαν κοινοτικά κονδύλια για την Άκουιλα η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου δεν θα πρέπει να συζητηθεί μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στην Ιταλική Βουλή. Και ερωτώ αν έγινε κάτι τέτοιο. Η έκθεση αναφέρει ότι τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν ήταν 150%, κάλυπταν 150% των τιμών αγοράς. Από τα 500 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, 350 εκατομμύρια αξιοποιήθηκαν για άλλους στόχους από αυτούς που είχαν προσημειωθεί ή από αυτό που είχε εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρησιμοποιήθηκαν για μόνιμες κατοικίες, αντί για προσωρινές, για παράδειγμα. με αποτέλεσμα να κατασκευαστούν πολύ λιγότερες κατοικίες από, από ό,τι αρχικά είχε προβλεφθεί και για τον λόγο που είχε δοθεί και η σχετική έγκριση και τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έπρεπε τα κονδύλια αυτά να είχαν αξιοποιηθεί πολύ περισσότερο στην Ιταλία. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ή ένα πάθημα κατά κάποιο τρόπο που θα μπορούσε να μας γίνει μάθημα, ώστε να κάνουμε κάποιες αλλαγές στο μέλλον. Ερωτώ λοιπόν, η ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου για την Άκουιλα συζητήθηκε στην Ιταλική Βουλή και αν ναι, ποια συμπεράσματα αντιλήθηκαν από αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Έχω άλλους δύο συναδέλφους. Ένας συνάδελφος από το Κροατικό Κοινοβούλιο, κύριος Διόκοβιτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Καλντέιρα, τον πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου, για την ε, εκτενή του παρουσίαση της ε, γνώμης του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ήταν πολύ σημαντικές οι προτάσεις που μας έκανε και θα μπορούσαμε να αντλήσουμε και πολλά συμπεράσματα από αυτές. Γιατί η αποτελεσματικότητα μπορεί να ελεγχθεί μόνο εφόσον έχει γίνει σωστή προετοιμασία. γιατί η προετοιμασία είναι θεμελιώδες ε, ε, τμήμα της επιτυχίας και της σωστής αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων. Γι' αυτό η σημερινή συζήτηση για μας ε, έχει ανεκτήμητη σημασία, όχι μόνο για να αποφύγουμε λάθη, αλλά και για να αξιοποιήσουμε καλύτερα και πιο ποιοτικά τα κοινοτικά κονδύλια. Φυσικά, περισσότερη έμφαση θα πρέπει να δώσουμε στην αποτελεσματικότητα και στη σωστή αξιοποίηση των κονδύλιων. Η σωστή λοιπόν προετοιμασία και ο έλεγχος της προετοιμασίας θα έχουν ε, κεφαλαιόδη σημασία για την έγκριση αυτών των κονδυλίων. Και φυσικά ο έλεγχος ε, της εκτέλεσης των κονδυλίων επίσης είναι σημαντικός. Γιατί από τη στιγμή που ξοδευτούν τα κονδύλια, αν χάσουμε την ευκαιρία να ελέγξουμε την εκτέλεσή τους, τότε ερχόμαστε σε πολύ κακή θέση και ε, όπως μας είπε ο κύριος Κατέρα, το 4,8% που είναι το ποσοστό σφάλματος στην εκτέλεση του προπολογισμού δεν είναι καθόλου καλή επίδοση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε σε όλα τα προγράμματα και τα σχέδια να επικεντρωθούμε στην διαμόρφωση μέσω της κουλτούρας, να επιμορφώσουμε καλύτερα τους αρμοδίους, και σε φάση πρόληψη και προετοιμασίας ε, να επικεντρώσουμε τι προσπάθειες ώστε να έχουμε καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά του. Έτσι θα μπορέσουμε με πιο ποιοτικό τρόπο να αποφύγουμε τα προβλήματα και τα ποσοστά σφάλματος. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα με την καλύτερη κατάρτιση, με την καλύτερη επιμόρφωση και τη σωστή κουλτούρα. Γιατί η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων δεν έχει γίνει ακόμη ε, ε, τμήμα σημαντικό και για την πολιτική ελίτ. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει αυτή η κουλτούρα. Θα πρέπει να επικεντρώσουμε και τους πολιτικούς στην αξιοποίηση, στην αποτελεσματικότητα. Η υλοποίηση των αποτελεσμάτων είναι σημαντικό θέμα. Λοιπόν, συμφωνώ, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στη σωστή διαπαιδαγώγηση και στη σωστή προετοιμασία για να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που είπατε κύριε Κιούκοβιτς ανταποκρίνεται και αντιστοιχεί και στη δική μας πεποίθηση. Έχουμε κοινό συμφέρον. Και δεν είναι πάντα οι επιτροπές ελέγχου προϋπολογισμού ή ελέγχου το λογαριασμό που έχουν ε, μεγάλη προτεραιότητα στην πολιτική υψηλή θέση. Γιατί πολλοί ε, αισθάνονται άβολα όταν αυτά τα πράγματα συζητούνται δημόσια. Αλλά για να προχωρήσουμε θα πρέπει να διαμορφώσουμε μια συναντήληψη σε όλα τα κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι είναι ανάγκη να υπάρχει ένας δημοκρατικός έλεγχος του τρόπου με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα των φορολογουμένων. Και όταν γίνονται σφάλματα να αναλύονται και να ε, εξάγονται και συμπεράσματα. Αυτό ρώτησε και ο κύριος Σόντεγκαρτ. Ο συνάδελφος Κρογέρο. Καριέλο. Που θέλει να απαντήσει. Ζητώ λίγο την υπομονή σας που δίνω το λόγο στον συνάδελφο από την Ιταλία για να απαντήσει αμέσως στα ερωτήματα που του ετέθησαν. Sì, ehm, allora, la discussione in merito al rapporto... Μάλιστα. Η επί της ουσίας συζήτηση για την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου δεν έχει γίνει ακόμα στο δικό μας κοινοβούλιο. Όπως ήδη είπα στην προηγούμενη μου παρέμβαση, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε ως Επιτροπή Προϋπολογισμού την ε, διαθεσιμότητα για να προβούμε σε εις βάθος ανάλυση της έκθεσης και μάλιστα να κάνουμε και έρευνα για το ποια ήταν τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν σε αυτήν την χρήση και κυρίως να παρέχουμε στην Επιτροπή σας ε, τα στοιχεία για μια ευρύτερη ε, αξιολόγηση της υπόθεσης. Θεωρούμε ωστόσο πως είναι σημαντικό, σημαντικότερη η αρχή της διαφάνειας. Δεν υπάρχει νομίζω τίποτα για το οποίο να πρέπει να δικαιολογηθούμε, διότι ο στόχος είναι να δώσουμε ε, στέγαση στους σεισμοπαθείς επετέύθη. Άρα βέβαια αυτό πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο των κανόνων του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε έτοιμοι να δείξουμε με απόλυτη διαφάνεια τι, πόσα και πώς δαπανήθηκαν ε, από τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ένας αυστριακός συνάδελφος έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος είπε προηγουμένως ότι θα πρέπει να μειωθεί το διοικητικό άκτος ε, και ότι τα χρήματα πρέπει να πιάνουν τόπο. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απολύτως επί της ουσίας. Αλλά δεν είναι η μοναδική μέθοδος αυτή να ενισχυθούν οι έλεγχοι. Δηλαδή ε, θα πρέπει να ε, εφαρμόζονται σωστά ε, και να σχεδιάζονται σωστά ε, στοχευμένες στην πράξη οι οδηγίες και οι υποδείξεις, γιατί δεν συμβαίνει πάντα αυτό, πολύ συγκεκριμένα, ε, σε σχέση με το όσα λέγει το ελεγκτικό συνέδριο. Στην Ισπανία, Αυστρία και στην Πορτογαλία υπάρχουν κάποια οικόπεδα που θεωρήθηκαν δασικές εκτάσεις ε, ή πράσινο, αλλά είναι κυρίως βράχη και όχι δάσος και ομάλο έδαφος. Δεν είναι βοσκοτόπια. Υπάρχει ένας ε, μαθηματικός τύπος και μοντέλα σε υπολογιστές αλλά δεν είναι πολύ εύκολο να υπολογίσεις τώρα από όλα τα βοσκοτόπια ποια είναι τα οικόπεδα που είναι βραχώδη και ε, δεν αντιστοιχούν 100%. Χρειάζεται ένας απλός τρόπος να εξακολουθεί κανείς να μετράει ψηφιακά ε, ολόκληρο το έδαφος. Όταν είναι χορτολιβαδική έκταση κάτι και μια γελάδα ας πούμε περνάει όλο το καλοκαίρι στο λιβάδι, ε, να υπολογίζουμε ένα εκτάριο αναγελάδα και όχι να πηγαίνουμε να μετράμε την κάθε πέτρα. Αυτό δεν κοστίζει λεφτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσα ίσα κάνει οικονομίες και είναι εύκολο να ελέγχεται. Και ανταποκρίνεται και σε αυτά που ζήτησε ο πρόεδρος να μην είναι γραφειοκρατικές οι διαδικασίες και βαριές και τα λεφτά να δαπανώνται εκεί που χρειάζεται και με σωστό τρόπο στην οικονομία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ισελ. Από την Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών αγωνιστήκαμε πάρα πολύ σκληρά έτσι ώστε στο δημοσιονομικό κανονισμό να επιτευχθεί μια διοικητική απλούστευση. Ήταν η συγγήτρια η κυρία Γκρέσλε αλλά και οι σκιώδεις συγγητές και εγώ ως πρόεδρος στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο αγωνιστήκαμε πραγματικά και πρέπει να σας πω και επιτυχώς ε, στο τέλος να υπάρχει δυνατότητα έτσι καταποκοπής υπολογισμού και να μην ε, ε, ζητούμε ανάκτηση αμεληταίων ποσών. Είναι σωστό αυτό που είπατε όμως. Στο μέλλον στην νομοθεσία θα πρέπει να φροντίζουμε, να προσέχουμε τι γίνεται με την εφαρμογή για να είναι και πιο απλή. Διότι ένα τμήμα των λαθών εκεί παρατηρείται και το είδαμε και με τα μέλη ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου για το θέμα των δημοσίων συμβάσεων που κάνουν έκθεση αυτό τον καιρό και του ζητήσαμε να δούμε ε, μήπως χρειάζεται και έλεγχος των διοικητικών δαπανών για να συνυπολογιστεί σε αυτή την έκθεση. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε προς την κατεύθυνση αυτή, να μειωθούν δηλαδή τα ασφάλματα η κυρία Κρέσλε και οι άλλοι συνάδελφοι και εγώ είμαστε περίεργοι να δούμε τώρα πώς θα εφαρμόζεται αυτός ο δημοσιονομικός κανονισμός στην πράξη, στη διοίκηση των κρατών μελών αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνει πραγματικότητα αυτή η απλούστευση. Γι' αυτό θα παρακαλούσαμε τους συναδέλφους ε, να το κοιτάξουν αυτό. Στην εκτέλεση να ζητούν τα κράτη-μέλη να τους δίδουν και τα στοιχεία αυτά για τις διοικητικές δαπάνες ε, με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να είναι πραγματική απλούστευση και όχι να ανατρέπεται αυτό από κάποιες διοικητικές διατάξεις. Ε, άλλοι δύο συνάδελφοι ζητούν το λόγο. Δεν ξέρω κύριε Καλτέρα, θέλετε να μιλήσετε στο μεταξύ μετά τους δύο συναδέλφους, ίσως να απαντήσετε. από την Τσεχική Γερουσία. Η κυρία Ντάγμαρ Τσβερίνοβα, παρακαλώ. Dobrý den, vážení kolegové, kolegyně. Dovolte, abych také za Českou republiku zde něco... Κυρίες Kyrie, να πω δύο λόγια εξ ονόματος ε, της τσεχικής ε, δημοκρατίας που αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόνο ένα ε, σώμα, το η Γερουσία, διότι το δεύτερο σώμα ε, βρίσκεται στη συντακτική του, συστατική του μάλλον διαδικασία και γι' αυτό και έρχεται μόνο εκπροσώπους της Γερουσίας της τσεχικής δημοκρατίας εδώ. Είχαμε κάποια προβλήματα όσον αφορά την χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και μάλιστα υπήρξαν και κάποια σφάλματα γιατί η δομή που δημιουργήθηκε ήταν εξαιρετικά περίπλοκη και στη συνέχεια ήταν δύσκολο να εφαρμόσουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ε, είναι ένα μεγάλο δίδαγμα για το μέλλον. Ε, να ευχαριστήσω δε τον ε, προλαλήσατε από την Αυστρία, διότι κάποια προγράμματα και κάποιοι κανόνες είναι τόσο περίπλοκοι. Ίσως όχι για μας τους πολιτικούς, γιατί δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εφαρμογή των κανόνων αυτών στην πράξη, αλλά είμαστε το σώμα το οποίο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο τους. Στη συνέχεια όμως εφαρμόζονται οι κανόνες και εφαρμόζονται από ανθρώπους σε συγκεκριμένες τοποθεσίες και ορισμένε φορές οι κανόνες αυτοί είναι εξαιρετικά περίπλοκοι. Ίσως θα πρέπει να εκπαιδεύονται καλύτερα για να γνωρίζουν τι είναι αποδεκτό, τι όχι, τι πρέπει να ελεγχθεί και έπειτα, σε σχέση με κάποια προγράμματα, θα έπρεπε να έχουμε ε, πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί ορισμένα προγράμματα διαρκούν πολλά χρόνια και οι κανόνες ε, μπορεί να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ε, του Συμβουλίου. Το Τσεχικό Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει πολύ σοβαρά την κατάσταση και ε, γίνεται σοβαρή συζήτηση στο εθνικό επίπεδο. Θα θέλαμε λοιπόν να σας ζητήσουμε να υιοθετήσετε μια πιο ευέλικτη προσέγγιση σε σχέση με τα σφάλματα, διότι αυτά δεν είναι μόνο δικά μας σφάλματα, είναι κοινά σφάλματα, διότι διαχειριζόμαστε χρήματα ε, των ε, Ευρωπαίων φορολογούμενων και θα έπρεπε να μπορούμε να μοιραστούμε την εμπειρία και τις πληροφορίες σε σχέση με τα σφάλματα αυτά, ώστε να μπορούμε στο μέλλον να τα αποφύγουμε. Επίσης θα πρέπει το αποτέλεσμα να είναι πιο ορατό απέναντι στο κοινό, διότι το κοινό δεν γνωρίζει ότι ε, υπάρχει τέτοιος αντίκτυπος, το κοινό Γνωρίζει πως υπάρχει βέβαια κόστος, αλλά όχι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ίσως να γνωρίζει πόσες θέσεις δημιουργήθηκαν, ποιος αντίκτυπος υπήρξε για την απασχόληση, αλλά όχι ακριβώ τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και το πόσο αποτελεσματικά ε, ε, αποτελεσματικό ήταν το πρόγραμμα σε σχέση με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Γι' αυτό και θα ήταν πολύ θετικό να στοχεύσουμε καλύτερα με τα προγράμματα. Ε, γιατί κάποιες φορές τα προγράμματα που απαιτούνται από κάποια συγκεκριμένη περιφέρεια δεν αντιστοιχούν με το με τους στόχους που έχουν τεθεί και στη συνέχεια Πρέπει ο κόσμος να υιοθετήσει πιο ευέλικτες ε, προσεγγίσεις ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα. Οι όροι λοιπόν και οι συνθήκες θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένοι και ως προς αυτό θα πρέπει να ε, είμαστε σε θέση να ερχόμαστε πιο συχνά σε επαφή με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ja, vielen Dank. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο συνάδελφος Φανίγιου από τις κατοχώρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε θα ήθελα να επικεντρωθώ στη λογοδοσία και πάλι των ε, δαπανών των κοινοτικών κονδυλίων. Συμφωνώ με τον ε, Κροάτη συνάδελφο που είπε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις προϋποθέσεις που χρειάζεται. Όχι μόνο δηλαδή τα σφάλματα, αλλά τι χρειάζεται για να δαπανάτε σωστά ένα κονδύλι. Χρειαζόμαστε όμως και τις ε, πληροφορίες για τα ποσοστά σφαλμάτων. Είναι πολύ σημαντικό για να κάνουμε ε, συζητήσεις με νόημα στα Εθνικά Κοινοβούλια για το πώς να βελτιώνονται οι δαπάνες αυτών ε, των ταμείων από τα κράτη-μέλη. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καλντέιρα, εάν το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σε μελλοντικές του εκθέσεις προτίθεται να μας δίνει στοιχεία για τα ποσοστά ασφαλμάτων ε, ε, επιμερισμένα, ένα χώρα μέλος, όχι σε γενική αναφορά. Και τι κίνητρα θεωρεί πιθανά ή δυνατά για να βελτιωθεί η ε, λογοδοσία των μεμονωμένων κρατών μελών στη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Λοιπόν, έγιναν πολλές ερωτήσεις, εθίγησαν πολλές πτυχές που αναφέρονται στο έργο και στις εργασίες ε, του ελεγκτικού συναδρίου. Ιδιαίτερη συνάδελφος από την τσεχική δημοκρατία ρώτησε ποια υποστήριξη μπορεί να δοθεί από τα θεσμικά όργανα. Ίσως να μπορούσατε να απαντήσετε σε ένα πρώτο γύρο, κύριε Καλντέιρα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ε, ε, βουλευτές για τις ερωτήσεις τους. Ελπίζω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες με τις απαντήσεις. Πρόσφατα άκουσα την ίδια ερώτηση που ανέφερε ο βουλευτή από τι κάτω χώρε. Τι μπορούμε να κάνουμε για το ποσοστό σφάλματο των κρατών μελών. Είπα και στην άλλη επιτροπή ότι ο νέο δημοσιονομικό κανονισμό προβλέπει μια νέα βάση για την ε, δήλωση αξιοπιστία των ηθινόντων για την ε, χρήση των δημοσιονομικών κονδυλίων στα διάφορα επίπεδα. Ο νέος δημοσιονομικός ε, ε, κανονισμός προβλέπει μια ε, αλυσίδα δηλώσεων αξιοπιστίας. Η εθνική δηλώση αξιοπιστίας είναι η βάση και η τελευταίος κρίκος αλυσίδας είναι η συνολική δήλωση αξιοπιστίας της Επιτροπής. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε πρώτα σε εθνικό επίπεδο. Αν δίνονται οι σωστές πληροφορίες, ακριβείς πληροφορίες από το κράτος μέλος θα μπορέσουμε και εμείς να δώσουμε θετική δήλωση αξιοπιστίας. Εξαρτάται από τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από το κράτος μέλος και κατά πόσο αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αν λοιπόν έχουμε μια αποτελεσματική αλυσίδα δηλώσεων αξιοπιστίας θα έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο γιατί τα εθνικά κοινοβούλια θα έχουν έτσι και πολύ περισσότερες πληροφορίες, θα κατατοπίζονται καλύτερα για την αποτελεσματικότητα των φορέων διαχείρισης. Θα έχουν περισσότερα κίνητρα ώστε από την αρχή να προλάβουν ατασταλίες και παράτυπη κατανομή των κονδυλίων. Γιατί σήμερα, ανάλογα με τους τομείς βέβαια έχουμε διαφορές, σε μερικούς τομείς στα περιφερειακά κονδύλια, στα ταμεία συνοχής. Πάνω από το 50% των συναλλαγών που έχουμε ελέγξει το 2012 αφορούσαν περιπτώσεις όπου οι εθνικές διοικήσεις που ήταν αρμόδιες για τη διαχείριση αυτών των κονδυλίων και που είχαν στην κατοχή τους τις πληροφορίες που θα απέτρεπαν ατασταλίες δεν ανέλαβαν σωστά το ρόλο τους. Γιατί? Οπότε θα πρέπει αυτή την ερώτηση να τη θέσουμε στους ηθήνοντες ε, της διαχείρισης, στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει επίσης να γίνει μια καλύτερη ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο στην πιστοποίηση των εθνικών, αρχών διαχείρισης, των εθνικών φορέων διαχείρισης, καλύτερο έλεγχο και εποπτεία των ε, εθνικών ελεκτικών φορέων. Αλλά η, λύση, η πηγή είναι οι εθνικές αρχές. Ο κ. Καριέλο είπε πολύ σωστά ότι καλύτερη η πρόληψη από τη θεραπεία. Συμφωνούμε απόλυτα. Αν λοιπόν κατασκευάσουμε αυτήν την αλυσίδα αξιοπιστίας, δηλώσεων αξιοπιστίας με τέτοιο τρόπο, ώστε όλοι να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και τα κράτη-μέλη να δίνουν από την αρχή ακριβείς, συγκρίσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες, όλοι θα είμαστε σε θέση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε καλύτερη εποπτεία. Αλλά και σε εθνικό επίπεδο θα εξασφαλίζεται καλύτερη εποπτεία. Το να ζητάμε από το ελεκτικό συνέδριο να κάνει επίσης όρις έλεγχο των 28 χωρών μελών και να δίνει με ακρίβεια πληροφορίες υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος για κάθε κράτος δεν θα ήταν και πολύ αποτελεσματικό. Δεν είναι αυτός ο καλύτερος τρόπος ε, για να υλοποιήσουμε το στόχο μας. Για να είμαστε αποτελεσματικοί θα πρέπει από την αρχή, από τη βάση, να έχουμε ε, σωστά συστήματα χρηστής διαχείρισης και ελέγχου σε εθνικό επίπεδο. Είπαμε στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Αυστρία αναφέρθηκε ότι αυτό που προβλέπεται από το κράτος ως χορτονομή αφορούσε τελικά δάσος. Αλλά είναι δύσκολο να βρει το ελεκτικό συνέδριο πώς εντοπίζονται τα διάφορα αγροτεμάχια και τι καλύπτουν. Και αυτό το σύστημα μέχρι στιγμής δεν λειτουργεί. Αυτά τα θέματα είναι εθνική ευθύνη. Οι εθνικοί φορείς θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση. Δεν θα πρέπει να τα αφήνουμε όλα και να τα περιμένουμε όλα από τον ελεγκτή, από το ελεγκτικό συνέδριο. Ο ελεγκτής ε, ελέγχει το κατά πόσο η πραγματικότητα ε, αντικατοπτρίζεται, αντικατοπτρίζεται στα στοιχεία που δίνονται. Και έχουμε το σύστημα εντοπισμού των ε, τεμαχίων, των αγροτεμαχίων. Θα πρέπει να ξέρουμε τον προορισμό του κάθε τεμαχίου. Έτσι στο μέλλον θα αποφύγουμε τέτοια λάθη εσφαλμένου χαρακτηρισμού. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια ενημέρωση, σωστή επικαιροποίηση του συστήματος ε, εντοπισμού και χαρακτηρισμού των ε, τεμαχίων. Τώρα, είπαμε ότι θέλουμε να πλουστεύσουμε και να έχουμε μια πιο ελαστική προσέγγιση των σφαλμάτων. Πιστεύω ότι το θέμα των απλών κανόνων, των εύκολων, εύληπτων κανόνων που θα μας ευκολύνει και την εθνική διαχείριση και τον εθνικό έλεγχο, αλλά και την ευρωπαϊκή διαχείριση και τον ευρωπαϊκό έλεγχο. Πιστεύω ότι με τις νέες προτάσεις για τη νέα περίοδο προγραμματισμού χάσαμε μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Γιατί υπάρχουν πολλά επίπεδα νομοθεσίας, κάτι που περιπλέκει στο έπακρο το σύστημα και τη διαδικασία. Και μάλιστα ε, τα κράτη-μέλη θα προσθέσουν ένα ακόμη επίπεδο που θα καταστήσει ακόμη πιο περίπλοκη την όλη διαδικασία. Τώρα, τι προϋποθέσεις θα πρέπει ε, να ισχύουν για την καταβολή των κονδυλίων. Υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις για την επιλεξιμότητα που μερικές φορές είναι διαφορετικές στα κράτη-μέλη. Είναι που είναι το σύστημα από μόνο του περίπλοκο και τα κράτη-μέλη μερικές φορές επιτείνουν αυτήν την περιπλοκότητα προσθέτοντας νέες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Γι' αυτό και είπαμε στο ελεκτικό συνέδριο να προσανατολίσουμε την νομοθεσία στην επιδίωξη των αποτελεσμάτων και όχι μόνο στις ε, εισρωές και στην κατανομή των κονδυλίων. Συμφωνώ με τον κύριο Καμπρίτο ότι θα πρέπει να διερευνούμε την αποτελεσματικότητα της χρήσης των κονδυλίων. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε από την αρχή σαφείς στόχους. Ποιος είναι επιδιωκόμενος στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος, του συγκεκριμένου σχεδίου. Από τη στιγμή που είμαστε σαφείς για το στόχο, θα πρέπει να θεσπίσουμε και κατάλληλους δείκτες, ώστε να διευκολύνουμε και τους ε, αρμόδιους της διαχείρισης και του ελέγχου να κρίνουν κατά πόσο τα αποτελέσματα υλοποιήθηκαν. Και θέλουμε μεν προϋποθέσεις που θα σχετίζονται όμως με τα αποτελέσματα, όχι με τις ροές. Θα πρέπει οι πληρωμές να συνδέονται με τις συγκεκριμένες επιδόσεις των προγραμμάτων, με τα αποτελέσματα. Γιατί καλό είναι να κατασκευάζουμε ένα λιμάνι και αποθήκες και αποβάθρες, αλλά το θέμα είναι ε, το λιμάνι επιτελεί την αποστολή του και εξασφαλίζει μια σειρά υπηρεσιών και θέσεων απασχόλησης που χρειάζονται. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Όχι μόνο υποδομή. Και τα αποτελέσματα είναι σημαντικό κίνητρο για την καλύτερη τη διαχείριση. Γιατί τήρηση και συμμόρφωση με τους κανόνες είναι μία πτυχή, αλλά η υλοποίηση των αποτελεσμάτων είναι άλλη πτυχή, πολύ σημαντική. Θα πρέπει λοιπόν αυτά να τα προσέξουμε στον σχεδιασμό των προγραμμάτων, στον σχεδιασμό των στόχων, ήδη από την αρχή για να ξέρουμε τι ε, σκοπούς επιδιώκει κάθε πρόγραμμα. Θεωρώ ότι απάντησα στις ερωτήσεις. Θα ήθελα να πω στον κύριο Καριέλο ότι όντως το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο με ιδιαίτερη χαρά θα λάβει μέρος σε μια συζήτηση στην ε, Ιταλική Βουλή αν προσκληθεί για να παρουσιάσει την ειδική του έκθεση για την Άκουλα. Ο κύριος Ρούσο που είναι μέρος του Ελεκτικού Συνεδρίου παρουσίασε άλλες ε, εκθέσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου και είναι πολύ δραστήριος. Δεν είναι ο συγκεκριμένος συντάκτης της έκθεσης αλλά ο αρμόδιος ε, συνάδελφος του Ελεκτικού Συνεδρίου, πολύ ευχαρίστω θα έρθει στην Ιταλική Βουλή να σας παρουσιάσει την έκθεση. Άλλωστε, οι αιτήσει εκθέσει μα με βάση την συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποστέλλονται σε όλες τις εθνικές βουλές. Και όλες οι βουλές που ε, ενδιαφέρονται για τις ειδικέ εκθέσεις και που δεν στέλνονται συστηματικά στα Εθνικά Κοινοβούλια, μπορούν να, άμα στο ζητήσουν, να τις, να τις στείλουμε. Γιατί Έχουμε πάρα πολλές εκθέσεις, 25 και, και δεν ενδιαφέρουν όλες οι ειδικέ εκθέσεις, όλες τις εθνικές βουλές. Είναι σημαντικό, αν σας ενδιαφέρουν συγκεκριμένα στοιχεία, να μας το πείτε. Αλλά ο κύριος Χάιντερ μίλησε για μια νέα αρχιτεκτονική του ελεκτικού συστήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το σύστημα όμως θα πρέπει να το προσέξουμε από τα θεμέλια. Το κτίριο θα πρέπει να ξεκινήσει από τα θεμέλια και φυσικά να έχουμε στενότερη συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Ελεκτικοφορέων και του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, όπως κάνετε εσείς μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Δεν μπορούμε να έχουμε μια γενική εικόνα της κατάστασης αν δεν έχουμε στενή συνεργασία μεταξύ μας. Και κάτι τέτοιο υπερβαίνει το σημερινό θέμα. Ξεπερνάει τη συνοχή και την γεωργία. Αφορά το όλο σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης. Γιατί ακριβώς επειδή ισχύει η συναρμοδιότητα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για πολλούς τομείς. Τώρα θεσπίζουμε την ε, νέα Τραπεζική Ένωση με ενιαίο επεπτικό μηχανισμό, με ενιαίο κανονισμό για την εξηγήση των τραπεζών. Ποιος θα είναι εκεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Εθνικών Κοινοβουλίων, των Εθνικών Ελεκτικών Φορέων σε ό,τι αφορά την πτυχή της ε, εθνικής εποπτείας. Όλα αυτά τα ζητήματα θα μπορούμε να τα συναρθρώσουμε σε ένα ενιαίο σύστημα για να έχουμε μια πολύ πιο πιστή γενική εικόνα των ε, δημοσίων οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος στο λόγο είτε από τα Εθνικά Κοινοβούλια είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. δεν βλέπω κάποιον άλλον, οπότε θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Βακένα. Θέλει να κάνει κάποια καταληκτικά σχόλια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου συζητάται στο ε, κοινοβούλιο μας. Η κυρία Γουλμπακέιτε που ηγείται της Ανώτατης Αρχής Ελέγχου την έχει υποβάλει, παρουσιάσει στην Επιτροπή ελέγχου του προπολογισμού του Κοινοβουλίου μας και είμαστε πολύ ευτυχείς γιατί αυτό μας επιτρέπει να δούμε ποια είναι τα κοινά λάθη και ποια είναι τα δικά μας λάθη σε αυτό το πλαίσιο. Εμείς μπορούμε να αποκομίσουμε διδάγματα και με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουμε καλύτερο έλεγχο των δαπανών. Θα ήθελα να πω, βασιζόμενοι στην εμπειρία μας, ότι κάποιες φορές οι κανόνες μας είναι εξαιρετικά αυστηροί και είναι πολύ δύσκολο να τους εφαρμόσει κανείς για να μπορέσει μπορέσει να επιτύχει τον κύριο στόχο. Κάποιες φορές δηλαδή δεν καταφέρουμε να πετύχουμε τους κύριους στόχους λόγω των αυστηρών κανόνων. Θα έπρεπε ίσως λοιπόν να εξασφαλιστεί περισσότερη ευελιξία διότι τα προγράμματα τίθενται σε εφαρμογή και υλοποιούνται κατά τη διάρκεια 2-3 ετών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να επιτευχθεί ο στόχος και να μην χρησιμοποιείται μόνο απλά και μόνο το κονδύλι ε, πιστεύω πως όλοι μας, συμπεριλαμβανομένες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλες, όλα αυτά τα στοιχεία για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους. Ευχαριστώ. Ja, vielen Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σήμερα το πρωί ε, ανταλλάξαμε απόψεις και εμπειρίες πάρα πολύ εντατικά για τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται τα ε, κοινοβούλια των κρατών μελών αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι μπορούμε συνοψίζοντας να πούμε ότι αφενός είναι πάντα καλό να γίνονται τέτοιες ανταλλαγές ε, απόψεων γιατί πραγματικά Τώρα μαθαίνουμε ένας από τον άλλον και είναι καλό να ακούμε πώς μπορούμε να βελτιώνουμε την ίδια μας την εργασία. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει αυτή η καλή πρακτική και μάλιστα η βέλτιστη πρακτική να έρχεται στο προσκήνιο ε, εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου αλλά και έρευνες των Εθνικών Ελεκτικών ε, Συνεδρίων χρησιμοποιούνται όχι για να κατηγορηθεί κάποιος ή να το καθίσουμε στο εδόλιο του κατηγορουμένου, αλλά για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας όλοι για βελτιώσεις και για ε, καλύτερη διαχείριση και δεν μπορώ να, παρά να συμφωνήσω με τους συναδέλφους που είπαν προηγουμένως ότι τώρα που έχουμε τέτοια παγκόσμια χρηματοοικονομική και γενικότερη οικονομική κρίση και σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι τεράστιες και οικονομικές δυσκολίες είναι συγκεντρωμένη η προσοχή των πολιτών, ανδρών και γυναικών στον τρόπο με τον οποίο ε, χρησιμοποιούνται τα ε, χρήματα από τους φόρους που πληρώνουν. Νομίζω το είπε και ο συνάδελφος από τις κάτω χώρες. Η αποδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται και από αυτό. Να μπορούμε να αποδεικνύουμε ότι ο δημοκρατικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών είναι πάντα δεδομένο. Τουλάχιστον εμείς έτσι το ε, αντιλαμβανόμαστε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Επιτροπή ε, Ελέγχου και ευχαριστώ και τον κύριο Μπούλτερ που ε, μίλησε για τις ε, διαχειριστικές δηλώσεις των ε, κρατών μελών. Αυτό είναι πάγιο διακομματικό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Βάλκη και τον πρόεδρο Καλτέρα για τις προτάσεις τους και ευχαριστώ και εσάς εκπροσώπους των Επιτροπών Ελέγχων Προϋπολογισμών των Εθνικών Κοινοβουλίων και με χαρά σύντομα να συνεχίσουμε αυτή την αλλαγή. Και τώρα σας προσκαλούμε εδώ σε ένα, ένα γεύμα με σάντουιτς για να ε, έχουμε και την ευκαιρία διαπροσωπικών ε, συζητήσεων και διμερών επαφών. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στις Βρυξέλλες και ελπίζω να ήταν γόνιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων και να μπορέσουμε να τη συνεχίσουμε και στο μέλλον. Κυρίσω λοιπόν το πέρας της επίσημης ε, συνεδρίασης με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστώ πολύ.